Liebe Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η κοινή συνεδρίαση των τριών κοινοβουλευτικών επιτροπών προπολογισμών ελέγχου προπολογισμού και θεμελιωδών ελευθεριών. Περιμένουμε βέβαια τον πρόεδρο της Επιτροπής προπολογισμών, Άρχισα όμως για να μην χάσουμε χρόνο, διότι το πρόγραμμα είναι αρκετά αυστηρά δομημένο καταλήξαμε στην άποψη ότι είναι σημαντικό και οι τρει. Ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές που έχουν κοινά θέματα, για τα ταμεία δηλαδή, να συνέλθουν και να εξετάσουν τα ταμεία. Έχουμε πολλούς μηχανισμούς σε θέματα εξωτερικής πολιτικής με ε, λίγα χρήματα. Και γι' αυτό χαίρομαι που δέχτηκε και ο πρόεδρος Μωράης της Επιτροπής Θεμελιδών Ελευθεριών να συνεργαστεί. Έτσι λοιπόν, αφού σας απευθύνω και πάλι χαιρετισμό, να δώσω το μικρόφωνο αμέσω στον ε, συνάδελφό μου κύριο Μωράης. Αγαπητέ Κλοντ. Ευχαριστώ αγαπητή Ίγκε για τα λόγια καλωσορίσματος. Έχετε δίκιο, όπως συνήθως, σχετικά με τον αριθμό μηχανισμών, εργαλείων και την ανάγκη να τα χειριστούμε με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο και χαίρομαι που υπάρχει η προσέλευση συναδέλφων μας σήμερα και χαίρομαι που οι τρεις κοινοβουλευτικές μας επιτροπές συνεργάζονται. Γιατί άραγε είναι σημαντικό, διότι βέβαια για προφανεί λόγου άσυλο και μετανάστευση βρίσκονται υψηλά στην ημερήσια διάταξη μετά από την άρξη της κρίσης το 2015 και μόνο συγκεκριμένε λύσει μπορούν να δοθούν, εφόσον όμω αυτέ χρηματοδοτούνται από τον προπολογισμό. Μιλούμε λοιπόν για την υποδοχή μεγάλου αριθμού αφήξεων, που βεβαίω αυξάνουν ακόμα στην Ιταλία, ε, ενέργειε έρευνα και διάσωση στην Μεσόγειο ε, και ενίσχυση των ακτοφυλακών και συνοριαφυλακών, τα λεγόμενα hot spot, διότι έχουν ε, ήδη πολλές χιλιάδες ε, ανθρώπων που δέχονται εκεί. Όλα αυτά τα μέτρα στηρίζονται οικονομικά από τον προϋπολογισμό. Και σε ό,τι αφορά το διοικητικό προσωπικό που στέλνει ο ΕΑΣΟ ε, και στις χώρες μέλη. Έχει δημιουργηθεί και ένα έκτακτο ταμείο για να προσφέρει υποστήριξη για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανθρωπιστική βοήθεια δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, όσοι παρακολουθούμε στενά τα πράγματα αυτά γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στις ελληνικά νησιά εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιη για τα πρόσωπα που ζητούν άσυλο. Καλώ ήρθατε, κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή Υπολογισμών. Μόλι είπαμε ότι είναι σωστό που οι τρει κοινοβουλευτικέ επιτροπέ συνεργάζονται στενά. Οι ελληνικέ και οι ιταλικέ αρχέ καταγγέλουν την έλλειψη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια και οι μη κρατικές οργανώσεις και όσοι από εμά ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, τα γνωρίζουμε καλά αυτά, μα λένε ότι ο συντονισμό δεν είναι επαρκή, τα χρήματα έρχονται με πολύ καθυστέρηση και δεν υπάρχει επαρκή υποστήριξη. Και όσοι από εμά έχουν επισκεφθεί τα ελληνικά νησιά ή και την Ιταλία τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν η σημερινή ακρόαση ζητήθηκε από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ σε συμφωνία με τις άλλες δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές προϋπολογισμών και ελέγχου προϋπολογισμού για να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση, ποια πράγματα αποδίδουν και πού χρειάζονται βελτιώσεις για να εξασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός στο σύνολό του υποστηρίζει τις πολιτικές αυτές προτεραιότητες. Ευχαριστώ τις δύο άλλες συναρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για τη δέσμευσή τους για να αναζητηθούν απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές και για την κοινή διοργάνωση της ακρόασης. Έχω την τιμή τώρα να μπορώ να καλωσορίσω Θα έπρεπε να ερχόμαστε πάντα στην ώρα μα. Ε, δεν μιλώ βεβαίω για τον πρόεδρο τη Επιτροπή Περιπολογισμού, μιλώ για τον εαυτό μου, έτσι το ξεκαθαρίζω αυτό, γιατί και εγώ καθυστέρησα λίγο και δεν είχα δει ότι είναι ήδη παρούσα η Έμιλι Ορέιλι, που είναι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, ω γνωρίζετε όλοι και όλε, και η οποία έχει αντιμετωπίσει όλες τις σχετικές έρευνες, αλλά βέβαια και σε συνεργασία με τους εθνικούς διαμεσολαβητές έχει παρακολουθήσει όλες τις ε, εξελίξεις στο δράμα των ε, των μεταναστών και των προσώπων που ζητούν άσυλο. Χωρίς λοιπόν να μακρηγορήσω, θα ήθελα να δώσω το λόγο αμέσως στην ε, κυρία Ορέιλη για να αναλύσει την κατάσταση από την σκοπιά της. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την πρόσκληση που μου απευθύνατε για να μπορέσω να σας μιλήσω σήμερα η, αρχίζει η συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προπολισμό και είναι σαφέ, όπω λέχθηκε ήδη, ότι τα θέματα τη χρηματοδότηση των ζητημάτων μετανάστευση και προστασία εξωτερικών συνόρων θα είναι κέρια. Όχι μόνο για οικονομικού ε, λόγου, αλλά και για πολιτικού. Είναι γνωστό πόσο αμφισβητούμενη είναι η πολιτική μετανάστευση σε ολόκληρη την Ένωση. Θα ακούσουμε εμπειρογνώμονε σήμερα για το πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και με λογοδοσία σκοπός των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνεται να είναι διπλός. Να βελτιωθούν οι συνθήκες για τα πρόσωπα που ζητούν άσυλο με ειδική χρηματοδότηση και να μειωθούν οι πιέσεις στα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης, αυξάνοντας τον αριθμό των εξωτερικών συνοριοφυλάκων και του προεπολισμού του Frontex. Η στόχευση για ένα από τα μεγαλύτερα, μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αναγνώριση μιας πραγματικότητας που αλλάζει συνεχώς και γρήγορα. Συνδυασμός πολλών παραγόντων, αλλαγές κλίματος, εσωτερικοί εκτοπισμοί, δυνατότητες μετανάστευσης που ε, προσφέρουν νέες τεχνολογίες και η συνδεσιμότητα συνεχίζουν να κάνουν τη μετανάστευση να είναι ένα από τα κέρια θέματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε για πολλά χρόνια ακόμη. Όπως ε, σχολιάστηκε πρόσφατα, η μετανάστευση ανταγωνίζεται πλέον την, τα οικονομικά ως η, ο που οδηγεί τις ε, ε, δυτικές πολιτικές, τις πολιτικές της Δύσης. Σημαντικές προκλήσεις. Αυτές οι λεγόμενες μικτές ροές, η νέα δυναμική που προσφέρουν νέες τεχνολογίες, όλα αυτά καθιστούν την μετανάστευση δύσκολο θέμα και νομικά και πολιτικά είναι γνωστή η διαφωνία για την κατανομή βαρών και δύσκολη και στο ανθρωπιστικό επίπεδο γιατί οι άνθρωποι, οι πολίτες δηλαδή, βρίσκονται ανάμεσα στην προσωπική συμπάθεια για τα θύματα όπως το νεκρό παιδί στην παραλία και στην απώλεια πλέον του ατομικισμού όταν έρχονται οι μετανάστες με σε σημαντικές μάζες. Δεν είναι ξεχωριστά τα πράγματα αυτά τόσο καλά όπω έχει σχολιάσει ένα νομομαθή πανεπιστημιακό, θα θέλαμε στι νομικέ μα κατηγορίε. Σημαντικέ προκλήσει όμω για όλους τους Ευρωπαίους και για την κοινωνία που έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε. Και ακριβώς λόγω της ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο οικονομικά, αλλά λόγω και του ανθρωπιστικού χαρακτήρα που έχουν ακόμα ε, τα αξιακά μας συστήματα, ότι συνεχίζει να αποτελεί προορισμό επιλογής για πολλούς μετανάστες. Μεταξύ του 2014 και 2016, η μισή από τους συνολικά 6,7 εκατομμύρια ανθρώπους που ζήτησαν άσυλο καταχωρίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά πάντως περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν μπροστά από τις φυσικές καταστροφές και τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής από ότι ε, φεύγουν μπροστά από ε, εμφυλίους πολέμους και άλλες συγκρούσεις. Οι ροές αυτές γίνονται όλο και πιο καθαρές καθώς ανακατατάσσεται ο χάρτης σε όλη την γη των κατοικήσιμων περιοχών. Σύμφωνα με την έκθεση 2016, ακραίες συνθήκες ε, ε, του κλίματος θα οδηγήσουν σε μια μέση μετακίνηση 200 εκατομμυρίων ανθρώπων μέχρι το 2050 σε σύγκριση, ετησίως πάντα, σε σύγκριση με 25 εκατομμύρια σήμερα. Νέα, νέα λοιπόν γεγονότα τα οποία έχουν ληφθεί υπόψη για παράδειγμα σε πολλέ μεταναστευτικέ πολιτικέ, με ένα παράδειγμα τη νέα Ζηλανδία, που προσφέρει τώρα την ανθρωπιστική βίζα για ανθρώπου οι οποίοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τι αιστείε του στον ειρηνικό λόγο αλλαγή του κλίματο. Σημαντικέ πιέσει, λοιπόν και από την άλλη μεριά η ανάγκη προσέλκυση ανθρώπων με δεξιότητε για να στηρίξουν τι οικονομίε μα. Είναι ακόμα λοιπόν πιο σημαντικό τα χρήματα που στοχεύονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών να χρησιμοποιηθούν σωστά και να δοθούν κατάλληλοι πόροι, να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι και οι οργανισμοί για να βοηθήσουν με τη χορήγηση συμβουλών στη σωστή δαπάνηση των χρημάτων αυτών. Και χρειαζόμαστε ανθρώπους θα βοηθήσουν, διότι το κενό ανάμεσα στις κορνιζαρισμένες συνθήκες και ε, διακηρύξεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους τείχους των θεσμών μας, των θεσμικών μας οργάνων δηλαδή και η ε, πραγματικότητα απέχουν πάρα πολύ. Το να δοθεί στους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν μπροστά σε ακατανόμαστες διώξεις δεν είναι, ε, δηλαδή προστασία δηλαδή, δεν είναι εφάπαξ δράση δεν φτάνει να περάσουν στη, την Μεσόγειο και να του δοθεί ένα πρώτο γεύμα και κάποια ρούχα. Χρειάζεται πραγματική προστασία με πολλές περίπλοκες ε, δράσεις υποστήριξης σε πολλούς τομείς και μέσα σε, μια, σε, μια, κάθε μια χώρα μέλος αλλά και μεταξύ των χωρών μελών καθώς και η πολιτική εργασία να πιστεί ένας πληθυσμός που είναι διστακτικός ότι η αύξηση του αριθμού των ε, προσφύγων και μεταναστών δεν αποτελεί απειλή. Από την άλλη, από την πρακτική σκοπιά δηλαδή, το πώς θα χρησιμοποιηθεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι κάτι το οποίο ελέγχουμε εμείς. Ενώ δεν ελέγχουμε ας πούμε τις ε, θεομηνίες, ούτε τις φυσικές καταστροφές και τις κλιματικές αλλαγές. Για τους μετανάστες το να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει να φτάσουν στα εξωτερικά σύνορα. Και εδώ η, η Κομισιόν προτείνει να αυξηθεί ο αριθμό των συνοριοφυλάκων. Για να μην γίνει όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα διάφορο φρούριο, θα πρέπει να παρακολουθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το γραφείο μου έχει θέσει ερωτήσει σχετικά με τη συμμόρφωση με ανθρώπινα δικαιώματα του οργανισμού Frontex και έχει πραγματική καλή συνεργασία με τον οργανισμό αυτό. Οι περισσότερε από τι συστάσει μου για βελτίωση έγιναν δεκτέ Χάρη δε στην στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η μία σύστασή μου που δεν είχε γίνει δεκτή από τον Frontex, δηλαδή να δημιουργηθεί μηχανισμός καταγγελιών, εν τέλει έγινε δεκτή και αυτή. Όσο αυξάνει το μέγεθος του οργανισμού, τόσο πιο σημαντικό είναι το προσωπικό που απασχολεί να είναι ενήμερο των υποχρώσεων του που απορρέουν από τον χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων. Και αυτά τα παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά οι συνάδελφοί μου και εγώ. Ο μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό χειρισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει αύξηση τη χρηματοδότηση για μετανάστε, πρόσωπα που ζητούν άσυλο κλπ. Ωστόσο, αύξηση του επίπεδου των ε, ε, πόρων δεν αρκεί για να αντιμετωπιστούν όλες οι προκλήσει. Θα πρέπει να υπάρξει περισσότερο συντονισμό στο πολιτικό επίπεδο και μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικών οργάνων. Συνεργασία μπορεί να αυξηθεί και με την αυξημένη αλληλεγγύη μεταξύ χωρών μελών, παρόλο που υπάρχουν πολιτικές προκλήσει ε, ε, επ' αυτού. Εν ώψη όμως ελληπού επάρκειας αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μελών, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι και μέσα σε κάθε χώρα μέλο υπάρχουν φορείς όπως οι Ombudsman, οι Οργανισμοί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μη κρατικέ οργανώσει που μπορούν να προσφέρουν τεχνογνωσία και στήριξη για την σωστή κατανομή των πόρων και για τον συντονισμό με άλλους ε, συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γραφείο μου, για παράδειγμα, μαζί με 19 άλλους εθνικούς και περιφερειακούς ε, συνηγόρους του πολίτη, έχουμε εργαστεί από πολλά χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι οι αιτήσει που δεν γίνονται δεκτές επιστρέφονται σε τρίτη χώρα σε συνεργασία με τις χώρες μέλη και ότι οι άνθρωποι αυτοί δέχονται φροντίδα στη διάρκεια του ταξιδιού. Όμως για να μπορούν να δράσουν οι φορείς αυτοί πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στις λεπτομέρειες των ταμείων ασύλου, μετανάστευσης και ενσωμάτωσης. Και αυτά τα έχω φροντίσει ήδη από καιρού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σπρώχνοντας τις χώρες μέλη να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τα ταμεία ΑΜΙΦ. Μπορεί να γίνουν περισσότερα πράγματα ακόμα. Χρειάζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρε μέλη να προσέχουν την εκταμείευση των πόρων, ώστε και σε τοπικό επίπεδο να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αν χρησιμοποιούνται σωστά ή αν μπορούν ενδεχομένω να διοχετευτούν αλλού, ανάλογα με τι συνθήκε που αλλάζουν. Περισσότεροι διαθέσιμε πληροφορίε και για του εθνικού ε, ombudsmen αλλά και για άλλου χρειάζεται για να ελέγχεται ο τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται στι υποχρεώσει του οι χώρε μέλη, στι υπηρεσίε που προσφέρουν σε πρόσφατα που ζητούν άσυλο, χρησιμοποιώντας ε, τους πόρους του Ταμείου ΑΜΙΦ. Και χρειάζεται και, πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα, καθώ και επίση να δημοσιεύονται τα έγγραφα αυτά, ώστε να μπορούν οι αρμόδιοι να ανταποκρίνουν στα καθήκοντά του. Περισσότερε δημοσιευμένε πληροφορίε θα δώσουν και τη δυνατότητα να ελέγχονται οι ροέ των ευρωπαϊκών πόρων και ιδίω αν χρησιμοποιούνται σωστά, σύμφωνα με τις προτεραιότητες και στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίω και η ενσωμάτωση, η ένταξη είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σημαίνει ότι θα πρέπει τα πρόσωπα αυτά να έχουν στέγη και να μπορούν να ενταχθούν σε μια κοινότητα που πολύ συχνά είναι πάρα πολύ διαφορετική πολιτιστικά από αυτή που γνωρίζουν. Δεν μπορεί κανείς να είναι παρόν Διαρκώ εκεί. Είναι σημαντικό λοιπόν η ίδια η κοινότητα να εμπλέκεται στο έργο αυτό. Γιατί αν η σχέση αυτή δεν αποδώσει και δεν θα μπορέσει να αποδώσει τίποτε άλλο. Υπάρχουν και άλλε αποφάσει πάρα πολύ δύσκολε, σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση των προσώπων αυτών. Για την ώρα 80% σύρων προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνεργοι. Και αυτό δεν μπορεί να ισχύει μονάχα σε έλλειψη δεξιοτήτων ή σε έλλειψη γλωσσικών γνώσεων κλπ. Πρόσφατα το, το ε, περιοδικό Economist διερεύνησε το θέμα και βρήκε ότι κάποιες χώρες έχουν βρει πρακτικές λύσεις που δεν οδηγούν σε μείωση της απασχόλησης των τοπικών εργαζόμενων αλλά τους οδηγούν καμιά φορά και σε καλύτερες δουλειές. Σημείωσε ότι το να επιτραπεί στα πρόσωπα που ζητούν άσυλο να εργαστούν διευκολύνει την αποδοχή των μεταναστευτικών ρευμάτων. Το περιοδικό, μαγαζίν, ε, το περιοδικό συγγνώμη, Economist ε, κοίταξε το θέμα αυτό από οικονομική σκοπιά. Οι χώρες μέλη ωστόσο έχουν να ασχοληθούν και με άλλα θέματα, με τη διατήρηση αξιοπρέπειας του ατόμου και μια θετική αντιμετώπιση των ε, νεοεισελθόντων. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν φύλακοι, μικροί και μεγάλοι, τη βασική ανθρωπιά. Στην Ελλάδα πήγα έξω από την Αθήνα, βρήκα κέντρο υποδοχή μεταναστών οι ελληνικές αρχές δέχονται ότι είναι καλά διαχειριζόμενο ε, κέντρο διότι βρίσκεται κοντά στην ε, πρωτεύουσα. Παρ' όλα αυτά εξεπλάγει από την δέσμευση και από την μεγάλη προσπάθεια που κάνουν και οι ντόπιοι αλλά και οι αρχές για να διευκολύνουν τη ζωή των ε, προσφύγων και μεταναστών αλλά και να τους προσφέρουν ελπίδα. Σε πολλές χώρες απλοί άνθρωποι έχουν προσφέρει χείρα βοηθείας και χωρίς να τους ζητηθεί και έχουν προσφέρει βοήθεια στους ε, νεοαφιχθέντες στα χωριά και στις πόλεις τους. Με τους πιο απλούς τρόπους, με παροχή φαγητού, με συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, με την ε, προσέγγιση σε μικρά παιδιά, ώστε τα δύο μέρη των κοινοτήτων αυτών να μπορούν να συνεπάρξουν εποφελία και των δύο πλευρών. Χωρίς να θέλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ρομαντικοί ή ε, συναισθηματικοί για τα θέματα αυτά, γιατί οι ζωές των ανθρώπων δεν είναι ξεκάθαρα ε, δεν είναι τακτοποιημένες. Υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές και μάλιστα πολιτισμικές διαφορές οι οποίες οδηγούν σε βαθιές ανησυχίες και αγωνίες. Ωστόσο, χρειάζεται μια φωτισμένη και θαραλέα πολιτική ηγεσία η οποία θα δώσει, ή θα προσφέρει μια στέρεα δομή για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Δεν μπορεί καμιά χώρα μέλο να το κάνει μόνη τη, είτε μικρή, είτε μεγάλη, είτε φιλελεύθερη, είτε και λιγότερο φιλελεύθερη. Σε όλε τι χώρε αυτέ υπάρχουν άτομα και οργανώσεις στο κρατικό και στο μη κρατικό επίπεδο που έχουν τη διάθεση να συμβάλλουν στην πολύ δύσκολη δουλειά της δημιουργίας ενός πρακτικού φωτισμένου ανθρώπινου συστήματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των ανθρώπων αυτών που είχαν την ατυχία να μην γεννηθούν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Βράγλη για την ανακοίνωσή σας που μας υπενθυμίζεται κάποιες πραγματικότητες, κάποια καθήκοντα ανθρωπιστικά που έχουμε. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στο, στους από το γραφείο Μπρόγκελ για την παρουσίαση της πρόσφατης μελέτης με τίτλο «Τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, τις, ε, για τη μεταναστευτική πολιτική, την πολιτική ασύλου και ένταξης». Αυτή η μελέτη ανήκει στο φάκελο ε, των θεμάτων που θα εξεταστούν στην σημερινή ακρόαση. Έχουμε τους καθηγητές Ντάρβας και τον δόκτωρα Βόλφ. Έχετε και οι δύο το λόγο για 15 λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα κάνω την παρέμβασή μου στα αγγλικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας ζήτησε να κάνουμε αυτή τη μελέτη. Λέγομαι Βόλφ και σε λίγο θα δώσω το λόγο ε, στον κύριο Τβά, τον συνάδελφό μου, για να σας παρουσιάσει την μελέτη μας αυτή αυτή. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να πω εισαγωγικά είναι να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που κάνει, που διοργανώνει αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι ένας ε, συγκεκριμένος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε μια σύνθετη πραγματικότητα, μια σύνθετη πρόκληση, που είναι ε, μία από τις μείζονες ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών σήμερα, με βάση πολλές σφιγμομετρήσεις. Αυτό το θέμα, το θέμα της μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι ένα θέμα που θα πάψει να μας απασχολεί τα επόμενα χρόνια. Κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει ένα πολύ σημαντικό θέμα και τα επόμενα χρόνια και θα είναι πολύ σημαντικό και τις επόμενες δεκαετίες για τους Ευρωπαίους πολίτες, για πολύ απλούς λόγους. Ξέρουμε τι προκαλεί τη μετανάστευση, ξέρουμε ότι Υπάρχουν οικονομικοί λόγοι για την μετανάστευση, υπάρχουν δημογραφικοί λόγοι για τη μετανάστευση, αλλά φυσικά και οι πόλεμοι και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκαλούν μετανάστες. Αν κοιτάξετε λοιπόν τα οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία, βλέπετε ότι η γειτονική μας Ήπειρος, η Αφρική, είναι μία Ήπειρος όπου ζει πολύ έντονες δημογραφικές πιέσεις, ε, από ένα σε δύο εκατομμύρια θα διπλασιαστεί ο πληθυσμός της Αφρικής ε, τα επόμενα 30 χρόνια. Και παρά τους δεκάρικους λόγους που βγάζουμε στην ε, Ευρώπη, ότι έχουμε ας πούμε ένα σχέδιο για την Αφρική και ότι θέλουμε να, να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη Αφρικής για να μειώσουμε την μετανάστευση από εκεί, η πραγματικότητα ποια είναι. Καθώς θα βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση στην Αφρική, οι άνθρωποι θα θέλουν όλο και περισσότερο να μεταναστεύουν στην Ευρώπη από το αντίθετο. Γιατί, Γιατί θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν. Επομένω, οι πιέσει, οι μεταναστευτικέ πιέσει, κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθούν από την Αφρική. Τώρα, μα ζητήσατε να αξιολογήσουμε πολύ πιο συγκεκριμένα. Για να δω αν δουλεύει αυτό το μηχανάκι. Να αξιολογήσουμε λοιπόν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό και να σας δώσουμε μια ανάλυση, μια εποπτική εικόνα και μια αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων, ε, των Ενωσιακών Ταμείων για τη μεταναστευτική πολιτική και την πολιτική ασύλου και ένταξη. Θα ήθελα σας πω ευθύ εξ αρχή ότι δεν θέλουμε να ελέγξουμε τα ταμεία, δεν κάνουμε έλεγχο των ταμείων, δεν σας λέμε αν χρησιμοποιήθηκαν καλά ή άσχημα. Προσπαθούμε να κάνουμε μια επισκόπηση και μια ανάλυση ακαδημαϊκού τύπου ε, γιατί δεν έχουμε και πρόσβαση σε εμπιστευτικά στοιχεία. Θα θέλαμε επίσης να σας κάνουμε και κάποιες συστάσει για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη χρήση αυτών των ταμείων. Η μεθοδολογία μας βασίζεται στην ανάλυση ε, στοιχείων που είναι ανοιχτά στο κοινό, στο ευρύτερο κοινό. Από στοιχεία από συνεντεύξεις με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, ε, από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, από τη Frontex, ε, από το ΑΜΙΦ, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, αλλά και από συνεντεύξεις με διάφορους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με τις εθνικές αρχές, το Ισπανικό Υπουργείο, ας πούμε, το Ιταλικό Υπουργείο κτλ. Επίσης κάνουμε και μια μελέτη των ΜΚΟ, γιατί σε πολλές περιπτώσεις η ΜΚΟ είναι η τελική αποδέκτε των κονδυλίων των, Ευρωπαϊκών και Ενωσιακών Ταμείων. Και θέλαμε να ακούσουμε από αυτού ε, τι άποψη έχουν για τα κονδύλια αυτά και τη διαδικασία ε, Ωραία. Σας ανέφερα κάποια νούμερα για τη μετανάστευση. Του μετανάστες προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αριστερά βλέπετε ότι τα νούμερα αυξήθηκαν πάρα πολύ το 2015 και 2016 λόγω της μεγάλης αύξησης ετούν τον άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της κρίσης στη Συρία. Αλλά γενικά, αν κοιτάξετε τα νούμερα αυτά θα δείτε ότι το άσυλο δεν είναι ο βασικό λόγο ε, για να μεταναστεύσει κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, παραδείγματο χάρη το 2014, ο αριθμό μεταναστών που ήρθαν για οικονομικού λόγου ή άλλου λόγου, πέρα από το άσυλο είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνου που ήρθαν ε, αναζητώντα άσυλο. Τα νούμερα βέβαια μειώθηκαν μετά την ε, κρίση του 2015 και 2016, αλλά παρόλα αυτά είναι σημαντικά ψηλότερα από ό,τι ήταν πριν από αυτή την περίοδο και βλέπουμε μια νοδική τάση που ανάλογη με αυτή που σας είπα στην αρχή. Επίσης, τα νούμερα είναι αρκετά σημαντικά σε ό,τι αφορά την ενωσιακή μετανάστευση, που είναι τελείως διαφορετικό πράγμα, διαφορετικοί λόγοι. Να σας πω κάποια στοιχεία. Αυτή η μετανάστευση είναι η πράσινη γραμμή και δεξιά σας δείχνει τη μετανάστευση Ευρωπαίων πολιτών, πολιτών της Ένωσης, ε, εκτός των ανθρώπων που επιστρέφουν στη χώρα προέλευσής τους, έτσι. Ε, και βεβαίως βλέπετε τα νούμερα αυτά είναι λιγάκι μικρότερα από τα, τους μετανάστες που έρχονται από τρίτες χώρες. Τώρα, πού έχουμε φτάσει τώρα. Μετά από αυτή τη διαφάνεια θα πάρει το λόγο συναδελφός μου. Πού έχουμε φτάσει λοιπόν. Είμαστε στην εξή φάση. Τα σημερινά ποσά για τη μετανάστευση ε, αυξήθηκαν σημαντικά στο τρέχον πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η αρχική κατανομή ήταν 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ και τώρα έχουμε φτάσει στα 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μια αύξηση από 0,8% του πουδουπού στο 1,3% του τρέχοντος πουδουπού. Είναι σχετικά μικρό αυτό το ποσοστό του πουδουπού, αλλά η αύξηση ήταν αρκετά μεγάλη. Φυσικά αυτές είναι δαπάνες για τη μετανάστευση. Υπάρχουν και άλλες δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινωνικές δαπάνες κτλ. όπου τμήμα αυτών των χρημάτων πηγαίνει για τους μετανάστες. Αλλά δεν είναι δυνατόν να αναλύσουμε το στοιχείο αυτό χωριστά, γιατί δεν ξέρουμε αν τα ποσά αυτά χρησιμοποιούνται πραγματικά για μετανάστες ή για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο να σας πει τη συνέχεια. Κοιτάξαμε την κατανομή κονδυλίων αναχώρα και αναθέμα. Και αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι για τα δύο μεγαλύτερα ταμεία, το ΑΜΙΘ, δηλαδή το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η βασική κλίδα κατανομής αντικατοπτρίζει στοιχεία του παρελθόντος. Δηλαδή βασιζόμαστε στο μερίδιο των πολιτών τρίτων χωρών ε, στο συνολικό πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τα δεδομένα του 2010 και δεν αναλύσαμε το πώς άλλαξαν οι τάσεις αυτές. Ε, μάλλον όταν αναλύουμε τις τάσεις αυτές βλέπουμε ότι ε, έχουμε πολύ ουσιαστικές διαφορές. Επίσης, σε σχέση με τη βασική κατανομή υπάρχουν αυξήσεις στα κονδύλια, αλλά χρησιμοποιώντα την ίδια κλίδα κατανομή. Παραδείγματο χάρη, το Ηνωμένο Βασίλειο παίρνει τα, τη μερίδα του λέοντο. Ενώ δεν αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση. Ενώ η Γερμανία αντίθετα έλαβε πολύ λιγότερη χρηματοδότηση από το μερίδιό τη ε, σε μετανάστες. το μερίδιο της Ιταλίας ήταν ε, λίγο πολύ σωστό η Ιταλία και η Ελλάδα, θα ήθελα να τονίσω, λάβαν το μεγαλύτερο κομμάτι της κατεπίγουσας βοήθειας. Υπήρχε επιπλέον δηλαδή ε, βοήθεια που δεν βασίστηκε σε κάποιο συγκεκριμένο τύπο, αλλά σε ad hoc αποφάσεις. Πάντω, η βασική κλίδα κατανομής πρέπει να πω ότι είναι πολύ ξεπερασμένη, απαρχαιωμένη, πρέπει να αναθεωρηθεί και μάλιστα προτείνουμε στο επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο να μην αντικατορπίζει απλώ τα μεταναστευτικά στοιχεία του 2016-2017 ή οτιδήποτε ας πούμε στοιχεία έχετε στη διάθεσή σα, Ο τύπος θα πρέπει να μα επιτρέπει να κάνουμε αλλαγή σύντο χρόνο. Γιατί Μπορεί το 2025 ή το 2027, ας πούμε, άλλες χώρες να υποστούν μεγάλες μεταναστευτικές πιέσεις. Δεν θα σας πω πολλά για αυτή τη ε, διαφάνεια, απλώς εδώ έχουμε τεράστιες διαφορές. Η Ελλάδα ξοδεύει τα περισσότερα κονδύλια του ΑΜΙΦ για το άσυλο, η Πορτογαλία ξοδεύει τα περισσότερα για την ένταξη, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ξοδεύει τα περισσότερα κονδύλια του ΑΜΙΦ για επιστροφές. Οι χώρε θα πρέπει να έχουν κάποια ευελιξία βεβαίω για το πώ ε, χρησιμοποιούν αυτά τα κονδύλια, αλλά μια και αυτά τα κονδύλια υποτίθεται ότι θα πρέπει να εξυπηρετούν κοινού ευρωπαϊκού στόχου, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξαναδούμε το πώς ξοδεύονται αυτά τα κονδύλια. Το επόμενο βασικό σημείο είναι η εφαρμογή. Πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν έχουμε στην πραγματικότητα ουσιαστικά στοιχεία, καλά στοιχεία. Κοιτάμε διάφορα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθούμε να βρούμε διάφορα στοιχεία για την εφαρμογή και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε τι γίνεται για ε, το θέμα της εφαρμογής. Ε, έγιναν διάφορες μελέτες για το ΑΜΕΙΒ και το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε ανεπαρκή στοιχεία για την εφαρμογή. Αυτό που συλλέξαμε ε, ήταν κάποια στοιχεία για το σύνολο των 28 χωρών, αλλά εδώ στα αυτά τα νούμερα βλέπετε πόσο οι συνολικές Υποχρεώσει του 2014-2020 πόσο έχουν εκταμιευθεί. Και βλέπετε ότι το 6,2 6,2 ε, δισεκατομμύρια ευρώ ε, υποχρεώσεων έχουν γίνει και μόνο 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν πληρωθεί, έχουν πραγματικά εκταμιευθεί. Δηλαδή, οι πραγματικέ εκταμιεύσει δεν αντικατοπτρίζουν ενδεχομένω την εφαρμογή, γιατί μπορεί να συνεχίζεται η εφαρμογή, αλλά τα ποσά ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Πάντω, δείχνουν αυτά τα νούμερα ότι μόνο το 40% των υποχρεώσεων ε, των ε, πιστώσεων υποχρεώσεων έχουν πληρωθεί τα τρία, τα πρώτα χρόνια. Αυτό είναι ε, σοκαριστικό. Άρα η εφαρμογή καθυστερεί πάρα πολύ. Υπάρχουν δύο τρόποι επίσης να αξιολογήσουμε τα τρέχοντα ταμεία. Καταρχάς, είχαμε αρκετά μακροσκελής ε, συνεντεύξεις με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και εδώ σε αυτή τη διαφάνεια συνοψίζουμε έξι βασικά μηνύματα. Καταρχάς, πολλά, πολλοί ενδιαφερόμενοι φορείς παραδέχονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε έντονα στην πρόκληση μέσα στα όρια που της έδινε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έκανε ό,τι μπορούσε. Ήταν ίσως το περισσότερο που μπορούσε να κάνει αυτό. Αλλά απλώς ε, κάθε, κάποιες χώρες όπως στην Ελλάδα δεν υπήρχε το διοικητικό δυναμικό. Και αυτά τα μία πραγματικά βοήθησαν για να, για να καταφέρουν αυτές οι χώρες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θετικά στοιχεία, αλλά υπάρχουν και κάποια αρνητικά. Καταρχά, ο αριθμό των πολύ μάλλον φορεί ανέφεραν ότι το σύστημα το λογιστικό και το σύστημα το δημοσιονομικό είναι πολύ περίπλοκο. Ε, είναι πολύ δύσκολο να αυξηθούν οι χρηματοδοτήσει για οργανισμού. Κάποια κονδύλια ή κάποιοι τρόποι χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων δεν, δεν είναι αρκετοί, δεν είναι κατάλληλοι ας πούμε για τη χρηματοδότηση ή για περιπτώσεις κατεπίγουσες. Επίσης, ε, διάφορες εθνικές αρχές ή ενωσιακοί οργανισμοί είπαν ότι υπάρχουν πολλές διοικητικέ δυσκολίες και διάφορες προποθέσει που παρεμποδίζουν τη σωστή εφαρμογή αυτών των ταμείων. Επίσης, ο συντονισμός, τεράστιο θέμα. Πολλές, σε πολλές συνεντεύξεις τονίστηκε ότι ο συντονισμός δεν είναι επαρκής. Ορισμένα θέματα εστιάζουν σε πιο τεχνικά σημεία, αλλά γενικά η έλλειψη συντονισμού ήταν ένα οριζόντιο θέμα. Το σημείο 4. Η τεράστια αύξηση της μετανάστευσης πίεσε πάρα πολύ, εφέρει στα ωριά του το προσωπικό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διάφορους οργανισμούς, ε, αλλά και σε εθνικές αρχές. Επίσης, είναι ασαφές πώς τα διάφορα ταμεία συνδέονται μεταξύ τους. Τι επικαλύψεις υπάρχουν, ποια είναι τα όρια δεν υπάρχει σαφή οριοθέτηση ανάμεσα στα διάφορα ταμεία. Χρειάζεται βελτίωση εδώ. Και τελευταίο και πολύ σημαντικό, σε πολλέ συνεντεύξει ακούσαμε ότι χρειάζονται περισσότερα λεφτά. Φυσικά. Η δεύτερη πηγή που χρησιμοποίησαμε ήταν η... χρησιμοποίησαμε αυτή την ε, μελέτη για τις ΜΚΟ. Μελέτη για 10 χώρες. Ε, κάναμε διάφορες ερωτήσεις, βέβαια δεν έχω πολύ χρόνο για να πω σε λεπτομέρειες, να σας τονίσω απλώς ότι αν συγκρίνουμε τα δύο βασικά ευρωπαϊκά ταμεία, το Κοινωνικό Ταμείο και το Αμύθ, το ΑΜΥΘ είναι πολύ πιο γραφειοκρατικό από το Κοινωνικό Ταμείο. Ενδιαφέρον αυτό. Και τα δύο ε, θεωρούνται πάντως πολύ γραφειοκρατικά σε σχέση με άλλα ταμεία που δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι είπαν ότι χρειάζεται καλύτερη, με απλούστευση για την καλύτερη χρήση αυτών των ταμείων. Θα πηδήξω διάφορες διαφάνειες και θα φτάσω στις συστάσεις. Πολύ γρήγορα. Όπως σας είπα ήδη, οι κλίδες κατανομής θα πρέπει να αλλάξουν. Ιδανικά θα πρέπει να έχουμε τύπους που θα επικαιροποιούνται από χρόνο σε χρόνο. Επίση, και μια και μεγαλύτερη προσθέμενη αξία ε, τη ευρωπαϊκή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης είναι ο συντονισμός των δράσεων των χωρών και για θέματα κατεπήγοντα. Θα προτείναμε λοιπόν να αυξήσουμε το μερίδιο της κατεπήγουσας βοήθειας και της ευελιξίας. Στην πρόταση που υπέβαλε στις 2 Μαΐου η Κομισιόν υπάρχει αύξηση όντω αυτή τη ευελιξία του προπολογισμού και τη δυνατότητα ανακατανομή για τη χρηματοδότηση του ΑΜΙΦ ή από το Σας είπα ότι χρησιμοποιείται για διαφορετικού σκοπού από χώρα σε χώρα και θα πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το θέμα. Φυσικά μπορούμε να κατανοήσουμε το πώ λειτουργούν αυτά τα ταμεία μόνο αν έχουμε καλά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε καλά στοιχεία, λεπτομερή στοιχεία για την εφαρμογή των διαφόρων ταμείων που αφορούν τη μετανάστευση. Πέντε. Πέμπτον, κάθε χώρα θα πρέπει να έχει μια ιστοσελίδα, απαιτείται αυτό, και να δημοσιεύει τις τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τα προγράμματα του ΑΜΙΦ. Εδώ βρήκαμε πάρα πολλέ ελλείψει σε σχέση με αυτήν την υποχρέωση και πολλέ χώρε έχουν πολύ παλιέ πληροφορίε και μάλιστα δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε αυτά τα στοιχεία. Επίση υπάρχουν πάρα πολλά άλλα ταμεία τα οποία δίνουν κάποια χρηματοδότηση για τη μετανάστευση, αλλά οι πίνακε δεν ήταν διαθέσιμοι δυστυχώ. Χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια, καλύτερα στοιχεία. 7. Ο δημοσιονομικός κανονισμός μερικές φορές εμποδίζει την σωστή εφαρμογή αυτών των ταμείων, τη σωστή χρήση αυτών των ταμείων. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, θα πρέπει να το ξαναδούμε. Το σημείο 8 είναι ο συντονισμός που είναι πρόβλημα, θα πρέπει να βελτιωθεί. Επίσης, ο αριθμός ε, των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε μονάδες όπου ασχολούνται με αυτά τα θέματα και αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση θα πρέπει να αυξηθεί. 10. Θα πρέπει να υπάρξει συνολική αύξηση χρηματοδότηση στο επόμενο πουδουπού Υπάρχουν σχετικές προτάσεις κομισιών, ε, εδώ και δύο εβδομάδε έγιναν, το, το σημείο 11. Οι, σκοποί των διαφόρων, οι στόχοι των διαφόρων ε, ταμείων θα πρέπει να διευκρινιστούν και οι επικαλύψεις να μειωθούν. Θέλουμε καλύτερες πληροφορίες και τέλος η ΜΚΟ μας έδωσαν διάφορες απαντήσεις. Τη συνοψίζω σε 15 παυλίτσες. Μερικές από αυτές είπαν ότι οι, πολλές φορές ε, μεγάλες ΜΚΟ παίρνουν πολλά λεφτά, ενώ δεν έχουν πρόσβαση επιτόπου, ας πούμε, ε, μέσω προσωπικού κτλ. Και άρα χρησιμοποιούν μικρότερες ΜΚΟ για να κάνουν τη δουλειά. Ε, επίσης, οι ΜΚΟ είπαν ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη άμεση ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ειδικά σε χώρες... Ε, που έχουν πρόβλημα για να υλοποιήσουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν και άλλες προτάσεις επίσης που θα ήθελα να εξετάσουν οι επιτροπές. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον καθηγητή Δραβές και τον συναδελφό σας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Ξέρω ότι εμ, εκτιμούμε όλα αυτά τα στοιχεία και τα γνωρίζουν φυσικά οι βουλευτέ τα στοιχεία αυτά, αλλά είναι καλό που μα τα παρουσιάσετε και με τον τρόπο αυτό. Ξέρω ότι έχουμε πάρε πολλέ ερωτήσει, αλλά θα προχωρήσουμε με την κυρία Μπεάτε γκαμίντερ από τη Γενική Διεύθυνση Home, που θα μας παρουσιάσει μια επισκόπηση της ε, τρέχουσας ε, νομοθεσίας και των δαπανών για την ε, μετανάστευση. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να σχολιάσετε και την έκθεση ε, Μπρίγκλ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τους Προέδρους και για τη δυνατότητα που μα δίνουν να βρισκόμαστε εδώ μαζί σα σήμερα και να παρουσιάσουμε και εμείς τη δική μας πλευρά. Και νομίζω ότι η χρονική συγκυρία της ακρόασης αυτής είναι πραγματικά πολύ επίκαιρη, γιατί είμαστε στη τελευταία φάση προετοιμασίας της ε, διάδοχης ε, νομοθεσίας για το ΑΜΙΦ και το ISF θα προταθεί στις αρχές Ιουνίου. Εξαιρετική λοιπόν η ευκαιρία που έχουμε να παρουσιάσουμε και εμείς από πλευρά της Επιτροπής τα τελευταία μας πορίσματα. Και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με την ε, μελέτη. Πολλές από τις συστάσεις μας συνάδουν με τη μελέτη, γιατί θεωρώ ότι και εμείς τα ίδια συμπεράσματα έχουμε καταλήξει και προφανώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές που εντοπίζουμε. Αλλά για να επανέλθουμε στην τρέχουσα κατάσταση. Είναι σαφέ. ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό σύστημα για το άσυλο. Αυτό παραμένει προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ανθεκτικοί σε μελλοντικέ κρίσει που θα ανακύψουν και να επιδείξουμε αλληλεγγύη και υπευθυνότητα ασφαλώ. Θα συνεχίσουμε να δείχνουμε αλληλεγγύη προ την Αφρική και να αντιμετωπίζουμε τη ρίζα τη μετανάστευση και να προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στι μακροπρόθεσμε προκλήσει. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτική μετανάστευση συμπληρώνονται και βαλτιώνονται όχι μόνο από τη χρηματοδότηση, αλλά με ε, σχέδια νομοθετικών πράξεων σε ό,τι αφορά το ε, κεφάλαιο, το, Ταμείο για την ε, Ενσωμάτωση και τη Μετανάστευση και το Ταμείο για την ιστορική Ασφάλεια. Άμυφ, λοιπόν, το Ταμείο για την Ενσωμάτωση και την Μετανάστευση υποστηρίζει διάφορες δράσεις όπως η νόμη μετανάστευση, η ενσωμάτωση, η ένταξη και ε, ασκήσεις επιστροφής. Το ISF, το Ταμείο αμα, για την Ιστορική Ασφάλεια, έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι ε, για την ε, βίζα, για τι θεωρήσει και το τμήμα της αστυνομίας για την ε, αστυνομική συνεργασία και για την ε, αποτροπή του νοριακού εγκλήματος. Όπως ήδη επισημάνθηκε, τα ποσά και εδώ βλέπω ότι είναι τόσο μικρά τα γράμματα που δεν τα βγάζονται προφανώς, ούτε εγώ τα βγάζω να σας πω την αλήθεια, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά όπως είπατε το τρέχον, ε, το τρέχον τα τρέχοντα κονδύλια έχουν αυξηθεί για τα επόμενα χρόνια και θα φτιάξουν το 10,8 ε, εκατομμύρια στο τέλη του 2017. Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα δαπανηθούν αυτοί οι πόροι. Και να σας πω ότι έχουμε τρεις τρόπους εφαρμογής και υλοποίησης των κονδυλίων αυτών. Κοινή ε, διαχείριση μεταξύ των κρατών μελών, άμεση διαχείριση όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εφαρμόζει τις δράσεις της Ένωσης και έμεση διαχείριση μέσω δηλαδή χρηματοδότηση διεθνών οργανισμών βάσει συμφωνιών που έχουν συναχθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι έχουμε μάθει λοιπόν ω τώρα, τι έχουμε διδαχθεί, γιατί το 2017 εξετάσαμε τα τρία χρόνια λειτουργία των διαταμείων του ΆΜΕΦ και του ISF, μαζί με τη νέα πρότασή μα ε, για τα διάδοχα ταμεία που θα συνοδευτούν από μία διάμεση ε, αναθεώρηση των δύο ταμείων. Τι έχουμε λοιπόν διδαχθεί, ποια είναι τα συμπεράσματα. Παρόμοια στοιχεία με αυτά που μας παρουσιάσατε και στην μελέτη σας. Τα ταμεία λοιπόν αυτά αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της κατάστασης που είναι πολύ δύσκολη. Έχουν καταδείξει την αξία τους και ως εργαλεία έκτητης ανάγκης αλλά και σε ό,τι αφορά μακροπρόθεσμη οικοδόμηση δυνατοτήτων και έχουν παίξει σημαντικό ρόλο τα τελευταία χρόνια για την βελτίωση των συστημάτων ασύλου και για την αύξηση των ικανοτήτων υποδοχής των κρατών μελών, προκειμένου να υπάρχει πιο ανθρώπινο περιβάλλον, πιο υγιές περιβάλλον κατά την άφηξη και την υποδοχή των ετών άσυλο. Υποστηρίζονται επίσης οι ευάλωτες ομάδες όπως η ε, ανήλικοι, οι ασυνοδοτοί ανήλικοι. Φτάνει λοιπόν και στα άτομα και στις οργανώσεις που έχει ως ε, στόχο για παράδειγμα, τα εθνικά προγράμματα του ΑΜΕΦ σε κοινή διαχείριση με τα κρατημέλη έχουν υποστηρίξει την υποδοχή πάνω από ένα εκατομμύριο του τον άσυλο. 160.000 εκ των οποίων ήταν ευάλωτα άτομα και ασυνοδευτεί ανήλικοι. Δημιουργήθηκαν πάνω από 60.000 ε, θέσει υποδοχές. Τετραπλασιάστηκαν δηλαδή σε σχέση με το 2014 οι εθνικέ αυτέ ε, θέσει ε, πολύ μεγάλο είναι και το προσωπικό το οποίο έχει καταρτιστεί και εκπαιδευτεί στις χώρες μέλη για την υποδοχή των ασύλων και πάνω από 33.000 άτομα έχουν επαναεκατασταθεί. Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι η παροχή αρρωγής προς τα, προς τα άτομα που έχουν ανάγκη η ενσωμάτωσή τους είναι σημαντικό σκέλος όλου του προγράμματος. 408.000 είναι οι δράσεις ενσωμάτωσης και ένταξης των ε, ετούντων άσυλο στα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, συγχρηματοδοτούνται και οι επιστροφέ. 127.000 άτομα επιστράφηκαν, ε, πολλά των οποίων επέστρεψαν θελούσια. Όπως αναφέρατε στα εθνικά προγράμματα, ε, μία από τις κριτικές ε, που ασκούνται, μία από τις επικρίσεις που ασκούνται, είναι ότι είναι αργή η απορρόφηση. Αυτό στέκει και δεν στέκει παράλληλα. Γιατί όταν ξεκινάει η προγραμματική περίοδο, προφανώ δαπανούμε κάποιο χρόνο στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό. Στη συνέχεια θα πρέπει προφανώ να εφαρμοστούν τα μέτρα, να υλοποιηθούν, να γίνουν κάποιε διαδικασίε, ε, διαγωνισμοί κτλ. Και μια και μιλάμε για λεφτά φορολογουμένων, θα πρέπει να ακολουθούμε του οικονομικού ε, κανόνε και να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και του Ευρωπαϊκού και του Εθνικού κανονισμού προφανώ. Γι' αυτό λοιπόν η απορρόφηση των πόρων μέχρι την πληρωμή μπορεί να πάρει χρόνο. Χρόνια, ολόκληρα. Γιατί προφανώ σε πρώτη φάση γίνεται ο σχεδιασμό, η υλοποίηση και μετά ξεκινά η εφαρμογή. Άρα ξεκινάμε με μια πρώτη χρηματοδότηση. Και μόνο προς το τέλος του προγράμματος ουσιαστικά λαμβάνουμε τις τελικές πληρωμές. Ως εκ τούτου, εξηγείται κάπως αυτό που κατέδειξε η μελέτη Μπρούγκελ, ότι στη φάση αυτή το 2017, γιατί μιλάμε για στοιχεία του 2017, η απορρόφηση ήταν μεταξύ 30 και 35% για τις πληρωμές. Θεωρώ ότι σε φάση αυτή είναι φυσιολογικό το ποσοστό αυτό. Άρα, εγώ να πω το εξή ότι είμαστε στη φάση κλεισίματο των λογαριασμών των κρατών μελών του 2017 και ήταν τεράστια η αύξηση για τα αιτήματα πληρωμών από τα κράτη-μέλη. Αυτό θα οδηγήσει προφανώ σε αύξηση των ποσοστών πληρωμών προ τα κράτη-μέλη από πλευρά τη Επιτροπή. Και τακτικά παρακολουθούμε το τι κάνουν τα κράτη-μέλη με τα χρήματα αυτά. Τα εθνικά προγράμματα τα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αλλαγέ προφανώ εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεργαζόμαστε με όλα τα κράτη-μέλη για να αξιοποιήσουμε τους πόρους που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και επίσης μόλις ολοκληρώθηκε η ενδιάμεση ε, αναθεώρηση για να δούμε πού ε, υπάρχει έλλειψη και που υπάρχει πλώνασμα πόρων. Γιατί σε κάποιε περιπτώσει δεν είναι ιδανική η κατανομή των πόρων και γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να εστιάσουμε τη χρηματοδότηση βάσει των καλύτερων δυνατών αξιών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον πολίτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα στοιχεία τα οποία επίσης ακούσαμε είναι το, το σύστημα ISF είναι πιο απλό από το σύστημα του AMIF, πιο εύκολο. Κοιτώντα ε, την κατάρτιση των ταμείων, πώς να συγκρίνουμε ένα πολύ νεαρό ταμείο, το ΆΜΙΦ του 2013, το οποίο λειτουργεί από το 2014, με ένα καταξιωμένο ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς διδασκόμαστε από αυτό και μαθαίνουμε. Είμαστε σε φάση προετοιμασίας της επόμενης γενιάς ε, ταμείων και προφανώς ε, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε όλες τις εμπειρίες που έχουμε συλλέξει από το παρελθόν. Τώρα, τι χρηματοδοτούμε πέρα από την κοινή διαχείριση έχουμε και το σκέλος της άμεσης διαχείρισης από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθείας μεταξύ 2014 και 2017 λεπτό. Έχουμε δαπανίσει 243 εκατομμύρια σε κινητικές δράσεις. 12 εκατομμύρια το 2014 μέχρι 140 εκατομμύρια πέρσι Αυξάνονται λοιπόν τα ποσοστά και κυρίως εστιαζόμαστε στην ε, μετανάστευση και στην ενσωμάτωση. Πρόκειται για επιδοτήσεις, ε, για ανοιχτές, ε, με ανοιχτούς διαγωνισμούς ή συγκεκριμένες συμφωνίες με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο IOM, το ECRE e κτλ. Επίσης έχουμε και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης. Σε αυτό το προπολογισμό σε, αυτά τα, σε τους πόρους. Και αυτό εγκρίνεται βάσει ετήσια ε, έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, έχουμε και στην εργαλειοθήκη μα ε, το εργαλείο έκτακτη ανάγκη. Το χρησιμοποίησαμε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των κρίσεων. Ένα οικονομικό το οποίο μα δίνει μια ευέλικτη δυνατότητα να παρέχουμε αρρωγή έκτακτη ανάγκη. Ε, με συγκεκριμένου όρου φυσικά. Συνήθω είναι ένα εφάπαξ ποσό το οποίο χορηγείται σε κράτη-μέλη, συχνά. 970 εκατομμύρια έχουν δαπανηθεί έτσι τα τελευταία τρία χρόνια. Βασικός ε, ε, δικαιούχος αυτών των πόρων τα τελευταία χρόνια ήταν η Ελλάδα. Το ανέφερε και ο κ. Μωράης. Έχουμε συνεργαστεί στενά. Έχουμε ένα οικονομικό σχέδιο για την Ελλάδα και με τις ελληνικές αρχές. Συζητιούνται όλα αυτά ε, άπαξ μηνιαίος Παρακολουθούμε σε πολύ ψηλό βαθμό επίπεδα την όλη διαδικασία στενά και η Ελλάδα έχει λάβει πάνω από 196 εκατομμύρια από το 2014 σε αρρωγή έκτακτης ανάγκης. Αυτό συγκεκριμένα για τις ελληνικές αρχές, για τη δημιουργία των hot spot και για την αύξηση των ικανοτήτων υποδοχών για να καλύπτουν και την υγειονομική περιθάλψη των μεταναστών. Επίσης, χρηματοδοτήσαμε 80 εκατομμύρια με την αρμοστία του ΟΗΕ για τη δημιουργία 80 εκατομμύρια λοιπόν δαπανήθηκαν μέσω του ΟΗΕ της αρμοστίας για τη δημιουργία θέσεων υποδοχή. Άλλες χώρες που έχουν ωφεληθεί είναι η Ιταλία και η Βουλγαρία. Η Ιταλία έχει λάβει πάνω από 190 εκατομμύρια και η Βουλγαρία πάνω από 170 εκατομμύρια σε τέτοιες ε, μη επιστρεπτές ενισχύσεις. Ε, νομική αρρωγή, λοιπόν, εντοπισμό των ευάλωτων ομάδων, αρρωγή για άτομα με συγκεκριμένες ανάγκες, κοινωνική βοήθεια, συγκεκριμένα μέτρα ε, και δράσεις επιτροφής ε, ενδεχομένω και άγορα υποδομών και υποκύποδομές και αγορά υλικού. Χρειάστηκαν λοιπόν τα χρήματα αυτά ιδιαίτερως κατά τη διάρκεια της κρίσης. Θα θέλαμε, ωστόσο, να μην χρειαζόμαστε διαρκώς ε, αρρωγή ε, έκτακτης ανάγκης. Είπαμε, είναι συγκεκριμένοι όροι. Και εργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη για να αυξήσουμε τις ικανότητες ανταπόκρισής τους με πιο διαφορετικό τρόπο, χρησιμοποιώντας κυρίως τα προγράμματα υπό τα εθνικά προγράμματα και την κοινή διαχείριση. Και τέλος, έχουμε και τις οργανώσεις που υποστηρίζουν το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην μετανάστευση, στον τομέα της μετανάστευσης. Κάποιες θα πάρουν και το λόγο λίγο αργότερα και προφανώς και αυτές λαμβάνουν χρηματοδότηση. Συνολικά, Θεωρώ ότι με το ΆΜΙΤ και το ISF και τα σχετικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τον εξωτερικό, τον κλάδο των εξωτερικών ε, συνεργασιών, αλλά και των ε, εσωτερικών εργαλειοθηκών. Έχουμε πολλά εργαλεία λοιπόν στη διαθέσή μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά φυσικά μόνοι μας. Πρόκειται για ένα συμπλήρωμα προφανώς σε σχέση με τους εθνικούς προπολογισμού και όσα προβλέπουν ως κονδύλια Παρ' όλα αυτά τα τελευταία τρία χρόνια της κρίσης ε, καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες υπό δύσκολες συνθήκες. Ευελιξία λοιπόν επέδειξε ο προπολογισμό και υποστήριξε σωστά την κατάσταση και έτσι πλέον νομίζω ότι μπορούμε να διδαχθούμε ε, για το μέλλον και να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα διδάγματα για την επόμενη ε, περίοδο του πολιτικού δημοσιονομικού πλησίου. Ευχαριστώ. Euh, Σας ευχαριστώ για τις ε, ενδιαφέρουσες διευκρινήσεις. Ως μαθαίνουμε από την ανακοίνωση, μα, από την, από την ε, ε, που προηγουμένως, θα αρχίσουμε το πρώτο πάνελ, το οποίο θα διευθύνω εγώ μαζί με τον συνάδελφό μου Κλοντ Μωράης. Το οποίο πρώτο πάνελ έχει ως τίτλο από την ε, διάθεση μέχρι την εφαρμογή. Για το Ταμείο ε, Ασύλου και Μετανάστευσης και το πάνελ αυτό έχει ως στόχο την πρώτη φάση του δημοσιονομικού κύκλου. Θα μας επιτρέψει να παρακολουθήσουμε τις ροές ε, των κονδυλίων από την στιγμή που θεσπίζονται οι στόχοι στο πολιτικό επίπεδο μέχρι την κατανομή των ε, κονδυλίων και μέχρι την υλοποίηση των έργων επιτόπου. Θα ακούσουμε τις ε, εμπειρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι συνεργάτες μας επιτόπου και οι προγνώμονες για τη, μετα... για τη μετανάστευση. Πρώτα λοιπόν το λόγο θα παραδώσω στον ε, συναδελφό μου κύριο Μωράης. Ευχαριστώ Ζαν. Πραγματικά είναι θαυμάσια τα μέλη που συναπαρτίζουν το πάνελ σήμερα ο Γιώργος Καμίνης, ήμαχος των Αθηναίων, ο οποίος θα λάβει τον λόγο και βέβαια και στη συνεργασία για, τον, για την ενσωμάτωση μεταναστών και προσώπων που ζητούν άσυλο. Και ο κ. Λετζέρη, Φαμπρίς Λετζέρη, εκτελεστικός διευθυντής του Frontex, ο κ. Ζαν Πιέρ Σεμπερί, επικεφαλής της επικοινωνίας η Ζωζεφίν Λίβελ της, ε, της International Advocacy και η Δόκτωρ Λίλιαν Σέρντι του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Για να κρατήσουμε λίγο και τον χρόνο μας, βεβαίως γνωρίζω ότι και οι ευρωβουλευτές έχουν ερωτήσεις που θα ήθελαν να υποβάλουν αυτός άλλωστε είναι ο στόχος της σημερινής ε, συζητήσεως, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τηρήσετε ένα χρονικό όριο παρεμβάσεως 8 λεπτών. Γιατί ξέρω ότι θα έχετε να απαντήσετε και ερωτήσεις από τα μέλη μας. Θερμό καλώς ορίσατε στον Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων. Παρακαλώ λάβετε το λόγο. Thank you, Mr. Chairman. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, αγαπητοί Πρόεδροι των Επιτροπών, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση σε αυτή την κοινή ακρόαση καθώς μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Κατά την περίοδο 2015-2016, με το πέρασμα εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων από την πόλη μας, βρεθήκαμε σε μια εξαιρετικά επίγουσα κατάσταση. Έπρεπε να προχωρήσουμε γρήγορα και με σχέδιο, καθώς και να βρούμε πόρους. Σήμερα, δυόμιση χρόνια μετά, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα πως η Αθήνα δεν θα είχε διαχειριστεί σωστά την προσφυγική κρίση χωρίς συνέργειες με ευρωπαϊκούς εταίρους και χωρίς πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους. Στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων η Αθήνα διαχειρίζεται συνολικά πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ για θέματα μεταναστών και προσφύγων. Πόροι που μας επιτρέπουν να διασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους πρόσφυγες, να προσφέρουμε πρόσβαση σε έγκυρη πληροφόρηση, να συντονίσουμε πάνω από 75 μη κυβερνητικέ οργανώσεις και κρατικούς φορείς, να δοκιμάζουμε νέα καινοτόμα προγράμματα κοινωνικής ένταξης. Όλα αυτά χωρίς την παραμικρή ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Από την αρχή της κρίσης προσπαθήσαμε να βρούμε πόρους όπου και αν αυτοί ήταν διαθέσιμοι. Η Αθήνα ήταν η πρώτη ελληνική πόλη που διεκδίκησε πόρους από το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ. Στη συνέχεια ακολούθησαν και 13 δήμοι σε όλη τη χώρα που συνέβαλαν καθοριστικά στην διαχείριση της κρίσης. Μέσω του προγράμματος αυτού έχουμε καταφέρει να στεγάσουμε έως σήμερα σε 300 διαμερίσματα στην πόλη πάνω από 4.000 άτομα. Συναντήσαμε όμως και εμπόδια, καθώς η νομοθεσία δεν είχε προβλέψει απορρόφηση κονδυλίων από δημοτικές αρχές. Δυστυχώς τα εμπόδια αυτά προκάλεσαν καθυστέρηση τουλάχιστον τριών μηνών στην έναρξη του προγράμματος. Βρήκαμε χρήματα για τη δημιουργία κέντρων ένταξης μεταναστών μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Συμμετείχαμε στο πρόγραμμα Αστικές Καινοτόμες Δράσεις, το Urban Innovative Actions, και πετύχαμε την έγκριση ενός πιλωτικού προγράμματος με την ενίσχυση 5 εκατομμυρίων ευρώ για να δοκιμάσουμε ένα καινοτόμο μοντέλο κοινωνικής ένταξης καταφέραμε να πάρουμε χρηματοδότηση ακριβώς επειδή το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά σε δημοτικές αρχές. Θέλω επίσης να σταθώ εδώ σε δύο πολύ χρήσιμα προγράμματα που εμείς οι ίδιοι εκπονήσαμε. Αναφέρομαι σε αυτά γιατί η ιστορία τους είναι νομίζω αποκαλυπτική για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις στην χρηματοδότηση. Μιλάω για ένα κέντρο συντονισμού που δημιουργήσαμε για 75 οργανώσεις και υπηρεσίες στην πόλη καθώς και το παρατηρητήριο προσφυγικών ροών που μας έδωσε πολύ σημαντικά στοιχεία σχετικά με τα θέματα ένταξης. Και τα δύο προγράμματα τα καταθέσαμε ως απολύτως επεξεργασμένες και κοστολογημένες προτάσεις μόλις ανακοινώθηκε το ΑΜΕΦ. Δυστυχώς, το αρμόδιο Υπουργείο λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων δεν μπόρεσε να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να προχωρήσουν. Τα προγράμματα υιοθετήθηκαν πάντως αμέσως από φιλανθρωπικά ιδιωτικά ιδρύματα και σήμερα θεωρούνται από τα πιο επιτυχημένα. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, η ιδιωτική επιχορήγηση έχει ημερομηνία λήξεως. Κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να σας μιλήσω μόνο για τη δουλειά που έχουμε κάνει στον Δήμο της Αθήνας και τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει. Σήμερα, εκ μέρους και του Partnership for the Inclusion of Migrants and Refugees, θέλω να περάσω ένα πολύ σαφές μήνυμα διεκδικούμε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λειτουργήσουμε μαζί πιο αποτελεσματικά. Η εισήγηση που παρουσιάζω σήμερα είναι καρπός σημαντικής δουλειάς που έχει γίνει στο πλαίσιο του partnership και της urban agenda, της αστικής ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία δύο χρόνια με στόχο να τεθεί υπόψη όλων όσων συμμετέχουν στη συζήτηση με αντικείμενο το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027. Το συνολικό σχέδιο δράσης του Partnership αλλά και η συγκεκριμένη έκθεση συστάσεων που συζητάμε σήμερα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς αποτέλεσαν αντικείμενο διαβούλευσης και έγκρισης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης που εκπροσωπούνται στο Partnership, δηλαδή και από τα κράτη-μέλη. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Διαπιστώνουμε καταρχάς ότι ο σχεδιασμός για τη διάθεση των πόρων παραμένει αποκλειστικά σε επίπεδο περιφερειών και κρατών μελών. Οι πόλεις δεν συμμετέχουν σε κανένα στάδιο του σχεδιασμού, ενώ σε μερικά κράτη-μέλη οι τοπικές αρχές δεν αναγνωρίζονται καν ως επιλέξιμοι εταίροι. Επισημαίνουμε λοιπόν την ανάγκη για καλύτερη ευθυγράμμιση των ευρωπαϊκών πόρων με τις ανάγκες των τοπικών αρχών και την ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προτείνουμε επίση την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, περιφερειών και τοπικών αρχών, προκειμένου να προωθηθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ πόρων, ΑΜΙΦ, ERDF, ESF. Αυτό θα προσέφερε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων. Απόρρια των προβλημάτων στο σχεδιασμό είναι η περιορισμένη πρόσβαση των πόλεων στους πόρους, όπως θα αντιληφθήκατε από το παράδειγμα τη Αθήνα. Οι πόλεις χρειάζονται ευελιξία στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων και το πρόβλημα αυτό φάνηκε ξεκάθαρα κατά την προσφυγική κρίση της διετίας 2015-2016. Έχει όμως ανακύψει και σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών και ερικών. Γι' αυτό το λόγο προτείνεται από την έκθεση οι πόλεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να έχουν απευθείας πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους ταμείων όπως το ΑΜΥΦ. Προτείνεται επίση να διασφαλίζεται η πρόσβαση των τοπικών αρχών στου πόρου που τα κράτη-μέλη δεν απορροφούν. Η έκθεση περιλαμβάνει συγκεκριμένε συστάσει για τη δημιουργία μια ομάδα πιλωτικών πόλεων. Οι Δήμοι στρέφονται πλέον και στον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών με του οποίου συμπράττουν επιτυχώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτέ τι εξελίξει, δημιουργώντα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στην έκθεση υπάρχει πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμών ανάμειξης χρηματοδοτικών εργαλείων, financial blending facilities, για πόλεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα συνδυάζουν πόρους των ταμείων με δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τέλος, για να μην έχουμε μια αστική πολιτική δύο ταχυτήτων, αλλά και για να πετύχουμε συμπράξεις σε όλες τις κλίμακες, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί μέσω προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης η πρόσβαση και στις μικρότερες πόλεις που δεν έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Το ίδιο και για μη κυβερνητικέ οργανώσει. Τα συμπεράσματα αυτή τη σημαντική δουλειά τη σύμπραξη δεν οδηγούν σε ένα πλουστευτικό αίτημα των πόλεων για περισσότερα χρήματα. Εστιάζουν όχι σε περισσότερη αλλά σε αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση. Η Urban Agenda για εμά πρέπει να αποτελέσει μία από τι νέε παραμέτρου τη πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Τόσο οι μικρότερε πόλει όσο και οι πρωτεύουσε έχουν επανειλημμένα αποδείξει ότι έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις υπεύθυνα με στρατηγική και με συνέπεια. Και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω πως αυτό το μήνυμα έχει αρχίσει να διαχέεται σε όλη την Ευρώπη. Αναφέρομαι ειδικότερα στην πρόσφατη πρόταση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη χρηματοδότηση των τοπικών κοινοτήτων που υποδέχονται πρόσφυγες, προκειμένου πια να ξεπεραστεί η τοξική συζήτηση σχετικά με τις ποσοστώσεις υποδοχής ανάμεσα στις χώρες. Οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται συνεχώς και σε αυτές προτίθενται οι δευτερογενείς μετακινήσεις. Οι πόλεις δέχονται μεγάλες πιέσεις. Απαιτείται μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα πρώτης υποδοχής και ένταξης, καθώς και η αντιστοιχή χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank uh, Ο πρόεδρος Κλοντ Μωράης. Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Καμίνη, και που κράτησε κιόλα το, τήρησε το χρονικό όριο. Θαυμάσιο αυτό, διότι θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε με κάποια ταχύτητα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Έχουμε τώρα τον δόκτωρα Λετζέρη, βεβαίως διευθυντή της Frontex, του Frontex. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών και εσείς κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Προϋπολογισμών και εσείς κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Οργανισμό Φύλαξης Συνόρων και Ακτών που έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην κοινή αυτή συνεδρίαση. Η δική μου παρέμβαση θα αναφερθεί στις δαπάνες που καλύπτουν το θέμα της προστασίας των συνόρων τίτλο. Θα ήθελα να αναφέρω προκαταρκτικά κάποια δεδομένα για τον προπολογισμό του Frontex και την εξέλιξή του από τη νέα του εντολή ως Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ακτοφυλακής και Συνοριαφής. Το 2018 320 εκατομμύρια και το 2019 προβλέπεται να είναι 333 εκατομμύρια ευρώ. Στον προπολογισμό βεβαίω υπάρχουν διάφορε κατηγορίε στον προπολογισμό του οργανισμού μα. Μπορεί όμω ήδη κανεί, οι δικαιούχοι των δαπανών που πληρώνει δηλαδή ο οργανισμός στη μεγάλη του πλειοψηφία είναι εθνικές υπηρεσίε των χωρών μελών οι οποίες συνεισφέρουν ε, των δαπανών εξοπλισμού διότι οι συμβάσεις, οι τρέχουσες συμβάσεις του οργανισμού που έχουν ως αποστολή την άβλωση, μίστοση, η προμήθεια τεχνικού εξώσης οχημάτων φτάνουν σήμερα στα 45 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για συμβάσεις που τρέχουν. Και για το 2018 είναι της τάξης των 84 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιστροφή, δηλαδή για αυτό, ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώστε επίσης ότι η χρηματοδότηση του οργανισμού γίνεται από διάφορες πηγές. Βεβαίως, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δικαίωμα ψήφου εκτός ε, Δημοκρατία Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου που είναι εκτός Σέγγεν. Υπάρχει και χρηματοδότηση από χώρες μέλη που δεν είναι, είναι χώρες συνδεδεμένες με το Σέγγεν, ε, Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτερστάιν και υπάρχουν και πρόσθετες ή το πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης της Ανατολικής ε, Συνεργασίας, υπάτου για τα Δυτικά Βαλκάνια, ΑΦΙΚ, African Intelligence Community και σύντομα και η νότια συνεργασία. Πάλιο ερώτημα που συζητείτε σήμερα. Αξιολόγηση δηλαδή της αποτελεσματικότητας των δαπανών. Για να εντοπίσουμε τα αναγκαία διδάγματα και για την μελλοντική διαχείριση. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο σημαντικά σχίσματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και τα οποία συχνά μας εμποδίζουν από το να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικότερα τα κονδύλια. Το πρώτο ας πούμε σιλό είναι η διαχείριση των συνόρων όπως αντιτίθεται αυτή με την εσωτερική ασφάλεια. Τονίζω ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τη διαχείριση των συνόρων καθώς και οι επιχορηγήσεις του οργανισμού έχουν διτό σκοπό διαχείριση της μετανάστευσης και εσωτερική ασφάλεια, όπου συμπεριλαμβάνεται και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Με άλλα λόγια, επενδύοντας στον οργανισμό συμβάλλεται και στην εσωτερική ασφάλεια του χώρου ελεύθερης διακίνησης Schengen δεν μπορεί κανεί να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των δαπανών για τη διαχείριση των συνόρων εξετάζοντα μόνο την πτυχή της διαχείρισης της μετανάστευσης. Ε, παραπέρα όμως, η θαλάσσια πλευρά, γιατί είμαστε ακτοφυλακοί και συνοριοφυλακοί, είναι προφανές ότι έχουμε νέε αποστολέ που πρέπει να εκπληρώσουμε. Έχουμε στενή συνεργασία με άλλους θαλάσσιους φορείς τον Οργανισμό Ελέγχου Αλίας και τον ε, Οργανισμό Θαλάσσιας Ασφάλειας. Μαζί διαχειριζόμαστε σχετικές αποστολές. Συμβάλλουν και στην ασφάλεια, στην διαχείριση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα, μάλιστα συμβάλλουν και σε άλλες πολιτικές. Το δεύτερο ας πούμε σύνολο θεμάτων, ή αν θέλετε σιλό, το οποίο θέλω να αναφέρω εδώ, είναι ο οργανισμός και απέναντί του τα κράτη-μέλη. Παραδοσιακά έχουμε ξεχωρίσει τα πρώτα πρώην, ε, το Ταμείο ΑΕΣΕΦ και τα λοιπά, από τη χρηματοδότηση του οργανισμού. Είναι κατανοητό μεν να υπάρχουν δύο διαφορετικοί νομικοί μηχανισμοί για την ε, υποστήριξη που δίνουν οι χώρες μέλη. Οφείλουμε ωστόσο να αντιληφθούμε την σημασία των συνεργειών και της ε, μεταξύ κρατών μελών και οργανισμού. Η νέα εντολή του οργανισμού λέει ότι η διαχείριση, και η φύλαξη των συνόρων είναι κοινή αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής, συντρέχουσα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκπροσωπείται εν προκειμένου από τον Frontex και των χωρών μελών. Δημιουργήσαμε πρώτα με τον κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοριαφυλακής, το, το Σώμα Συνοριοφυλάκων, συνεργασία εθνικών αρχών με τον οργανισμό, υπάρχουν και άλλα βέβαια παραδείγματα συνεργειών. Η ίδια στρατηγική στατική ανάλυση του οργανισμού και ιδίω η αξιολόγηση τροτότητας, που συναποτελεί μέρο τη νέα μα εντολή Και η νέα στρατηγική, η ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείριση των συνόρων, που θα πρέπει να εφαρμόσει ο οργανισμός από φέτος είναι η βάση για την οικονομική υποστήριξη των χωρών μελών. Μπορούμε δηλαδή εδώ να βρούμε τον αναγκαίο μηχανισμό για να κάνουμε μια στρατηγική ευθυγράμμιση και δημοσιονομική ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων μας. Τα προγράμματα συμπλήρωσης των διαφόρων πολιτικών και στρατηγικών και του οργανισμού και των χωρών μελών μας βοηθούν να αναπτύξουμε ικανότητες για να αντιμετωπίσουμε το ίδιο κοινό εξωτερικό σύνορο. Το ISF, Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, εξυπηρετεί τουλάχιστον στη θεωρία ως μηχανισμός που επιτρέπει την προμήθεια ε, βαρέως εξοπλισμού, όπως σκαφών, ελικοπτέρων κλπ. για τον οργανισμό. Έχω τώρα κάποια συμπεράσματα για το μέλλον θα ήθελα να συστήσω στην βάση των εμπειριών μας του Frontex δηλαδή, του Οργανισμού Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής, να γίνει ο σχεδιασμός στην βάση μιας μεθοδολογίας activity-based. Ποια είναι η συμβολή δηλαδή των διαφόρων ταμείων που έχουν πολλαπλούς σκοπούς, ώστε να έχουμε να, τη δυνατότητα ε, να ειχνηλατήσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κατανομή των κονδυλίων, αλλά και η λογοδοσία, ώστε από την άλλη μεριά να μπορούμε να ενημερώνουμε τα πρόσωπα που λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις για το τι γίνεται, ακόμα περισσότερο και πέραν από αυτά που έχουν ήδη ψηφίσει στις γραμμές του προϋπολισμού. Έχουμε δει και έχουμε υποστεί κιόλα τους περιορισμούς του διακυβερνητικού μοντέλου που αναζητεί αλλού πηγές χρηματοδότησης οι δεξαμενές προσωπικού και υλικού για τον ε, οργανισμό Frontex παραμένουν σε εθνική αρμοδιότητα και χρειάζεται εκεί να γίνονται διαπραγματεύσεις. Ούτε η προηγούμενη συνοριοφυλακή, ούτε και τώρα οι συνοριοφυλακές δεν κατάφεραν να αυξήσουν τις εθνικές ικανότητες για να έχουν επαρκή εξοπλισμό για τις αποστολές Frontex. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και να διασφαλίσουμε ότι... Για ξαναπείτε αυτή την τελευταία φράση. Οι ίδιες ικανότητές μας, ό,τι αφορά υλικό εξοπλισμό δηλαδή και προσωπικό, για να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας, οι ίδιες ικανότητες δηλαδή του οργανισμού θα πρέπει να είναι η βάση για τις αποστολές μας, ενώ οι εθνικές συμβολές θα παραμείνουν συμπληρωματικές. Σύστασή μου για το μέλλον είναι ο μηχανισμός αλληλεγγύης των χωρών μελών, όπως προτείνεται στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα στρατηγικά κενά και να στοχεύσουν στον εξυγχρονισμό και καινοτομία. Επομένως, μέσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. οι επιχορηγήσεις να μας βοηθήσουν για να αντιμετωπίζουμε ιδίω περιπτώσεις κρίσεων, για να μπορούμε να αντιδρούμε ταχαίως. Και οι δύο μηχανισμοί χρηματοδότησης θα παρακολουθούνται λοιπόν προσεκτικά για το νέο χρηματοδοτικό μέσον και λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό του Frontex που εγκρίνεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος από την ΕΑΣΟ το πολύ πολύ 8 λεπτά. Ε, θέλω να ακούσουμε όλους τους ομιλητές του πάνελ, γιατί δυστυχώς, όπως γίνεται συνήθως, οι ευρωβουλευτές λίγο-λίγο φεύγουν, έχουμε διαρροές. Γι' αυτό σας παρακαλώ, θα ήθελα να ακούσουμε όλους τους ομιλητές. Έχετε το πολύ, πολύ 8 λεπτά. Μετά θα αναλάβει η συνάδελφος στην Προεδρία. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο που μας κάλεσε εδώ. Η κρίση του 2015 ανάγκασε την υπηρεσία μου την ΕΑΣΟ να αυξήσει τις ε, κατεπίγουσες επιχειρήσεις της. Ε, χρειάστηκε λοιπόν να υπάρξουν εκατοντάδες εμπειρογνώμονες και διερμηνείς για μας. Ε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν είχαμε καμία επιχειρησιακή δραστηριότητα μέχρι τότε μέχρι το 2015. Δεν είχαμε καμία εμπειρία λοιπόν. Επίσης δεν είχαμε και το διοικητικό υπόβαθρο που χρειάζεται για να υποστηρίξουμε τέτοιες επιχειρήσεις. Επιπλέον πολλές φορές η υπηρεσία χρειάζεται. Αν δεν ήμασταν εμείς θα τις είχαν καλύψει από τη χρηματοδότηση τα κράτη-μέλη του ΑΜΥΦ. Αλλά χρειάστηκε εμείς να παρέμβουμε. Παίξαμε ένα σημαντικό ρόλο, αλλά το χρειαστήκαμε επιπλέον κονδύλια και ήδη το 2015 ε, έγινε η πρώτη τροπολογία στον προπολογισμό και το 2000 κυρίως για την Ελλάδα και την Ιταλία και χρησιμοποιήθηκαν για να πάνε διερμηνείς, ε, εργαζόμενοι εκεί επιπλέον. Ε, επίσης για την Τουρκία χρειάστηκε επιπλέον χρηματοδότηση για τη συμφωνία με την Τουρκία και εδώ χρησιμοποίησαμε επίσης τις ΕΜΑ που τέσσερις φορές, Πρόεδρε. Πρέπει να το αναφέρω αυτό για να ανταποκριθούμε στις πολιτικές ανάγκες των ε, κρατών μελών. Και η ευρωπαϊκή συνεισφορά στον προπολογισμό της ΕΑΣΟ αυξήθηκε, εξαπλασιάστηκε ανάμεσα στο 2010, περνάει τα 92 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπετε την τρομακτική αλλαγή. Επίσης, μιλάμε για μια πρόταση που υπάρχει ε, για, το, για την ΕΑΣΟ, γιατί το ΕΑΣΟ θα αναλάβει και νέα καθήκοντα, τα οποία χρειάζονται βεβαίως επιπλέον χρηματοδότηση. Πιστεύουμε καθηκόντων της ε, ΕΑΣΟ και χρειαζόμαστε και την να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη, τα οποία δέχονται πιέσεις ε, λόγω αυξημένων ε, αναγκών στο επίπεδο του ασύλου. Αυτό το πρόβλημα θα παραμείνει και θα το αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον. Τι διδαχθήκαμε από το παρελθόν. Καταρχάς, η ικανότητά μας να κινητοποιούμε γρήγορα κονδύλια, ειδικά για τους ε, οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί και να βελτιωθεί. Μάθαμε επίσης ότι οι δαπάνες μας, οι επιχειρηματικές μας δαπάνες, ε, είναι μόνο μερικώς προβλέψιμες. Δεν Επομένως, δεν μπορούμε να έχουμε μια προσέγγιση μονοκόμματη. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θα ήθελα να στείλω. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του ΑΜΙΦ, υποφεληθούν πολύ από υποστήριξη από την Κομισιόν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, γιατί μπορούν να τους διαθέσουν τεχνική πραγματογνωμοσύνη. Ε, για τη χρήση αυτών των κονδυλίων, αυτών των νέων από αυτά τα νέα ταμεία, από την εμπειρία μας σας λέω ότι πιστεύω ότι η χρήση των κονδυλίων αυτών από... Επίσης κάτι που το, όλοι το βλέπουν και κανένας δεν το συζητάει. Υπάρχουν τομείς όπου μπορεί να κάνει τη διαφορά η υπηρεσία μου. Παραδείγματο χάρη την οικονομική διαχείριση και τις ε, προμήθειες. Εκεί μπορεί να βοηθήσουμε. Παραδείγματο χάρη, ε, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο έκανε μια έκθεση και μια της ε, έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου του 2016 που οδήγησε στην απαλλαγή του προϋπολογισμού ε, για την επόμενη χρονιά. Καταλαβαίνουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, περιμένουμε την έρευνα που γίνεται από την Όλαφ για το θέμα αυτό της απαλλαγής. Θα σας πω καταληκτικά. Το πρώτο που θέλω να σας πω ότι η κρίση μας κατέλαβε εξαπίνης και εμάς στην ΕΑΣΟ ήμασταν απροετοίμαστοι. Δεν είχαμε την απαραίτητη εμπειρία τότε. Προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε όσο καλύτερα μπορούσαμε και πιστεύω ότι κάναμε τη διαφορά για την Ιταλία και για την Ελλάδα. Δημιουργήσαμε το πείσουμε τα του οίκου μας και να δώσουμε την υποστήριξη στα κράτη-μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πυρός, γιατί χρειάζονται αυτή την υποστήριξη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον επόμενο πανελίστα, την Ζουζεφίν Λίμπλ, από... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μιλώ εξ ονόματα στη ή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για του ε, Πρόσφυγε και τους εξόριστους. Ε, ε, μια ένωση 95 μοικείο για τον τομέα των, τον, τον και των μεταναστών και προσφύγων. Αυτά που δημοσιεύσαμε το Ιανουάριο του 2018. Στις αρχές λοιπόν του έτους. Και θα βασιστώ και σε στοιχεία των μελών του ECRE που χρησιμοποιούν η χρηματοδότηση του ECRE. Να κάνω μια ανακεφαλαίωση. Έχουμε άλλα τέσσερις ε, στόχους. Την ανάπτυξη, των σε ε, προτεραιότητα ασύλου, κατά εις δεύτερον ε, υποστήριξη της νόμιμης μετανάστευσης, βελτίωση δίκαιων στρατηγικών επιστροφών και αύξηση αλληλεγγύης και υπευθυνότητας και που ήδη αναφέρθηκαν λοιπόν. Αρχική ε, εκχώρηση των πόρων του ΑΜΙΦΕ για τα εθνικά προγράμματα και σε ό,τι αφορά την κατάσταση στις κρατές, στα κρατή-μέλη Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα. Έλαβαν τις πιο μεγάλες Αν δείτε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια τι γίνεται. Είναι σαφή λοιπόν που επίσης βλέπουμε και την αρρωγή έκτακτης ανάγκης στις διάφορες χώρες. Βουλγαρία, Ιταλία, βλέπετε στις χώρες αυτές όπου η ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για τους ε, διαμένοντες ε, τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους πρόσφυγες. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκχωρούν 20% της χρηματοδότησης στο άσυλο και 20% στις προτεραιότητες ένταξης και ενσωμάτωσης. Το πληρώνει πολύ μεγαλύτερο πολύ μεγαλύτερα ποσά για τις επιστροφές ε, πολύ μεγαλύτερο ποσό λοιπόν στις εκχωρήσεις και στο άσυλο. Αλλά η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε μεταξύ την εκχώρηση και της δαπάνης, της πραγματική ταπάνης, το επόμενο που το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης να περιλαμβάνει 15% ταμείο. Να δούμε τώρα τη διαφορά μεταξύ Έτσι υπάρχει μια συγκριτική επισκόπηση. Το ΆΜΕΦ λοιπόν σε γενικέ γραμμέ εφαρμόζονται και ακούσαμε και προηγουμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει αυτή η χρονοκαθυστέρηση ενών του Σεπτεμβρίου 2017. Βάση λοιπόν αυτό άλλωστε και αστυνομική βάση του Άμιφ ετήσιες εκθέσεις που προβλέπονται δράσεις από τους δικαιούχους και να ακολουθείται η γενική την υλοποίηση. Και άρα, για τη μελέτη αυτή καταρτήσαμε ένα ερωτηματολόγιο που το στείλαμε στις διάφορες υπηρεσίες που θέλουμε προφανώς να προαγάγουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συμπληρωματικότητα και η τελική προστιθέμενη αξία. Για... Ότι αντικαθιστά ουσιαστικά την εθνική χρηματοδότηση. Άρα στην επόμενη περίοδο θα πρέπει να κοιτάξουμε κατά πόσον όντω υπάρχει αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον επόμενο πανελίστα, την Dr. Ε, Λίλιαν Τσούρτη από το δίκτυο Οδυσσέας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ε, ευγενική σας πρόσκληση και είμαι τελευταία ομιλήτρια, αν δεν κάνω λάθος. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και να είμαι και συγκεκριμένη. Αν υπάρχει λοιπόν ένα βασικό μήνυμα για τη μεταρρύθμιση των ταμείων είναι να απομακρυνθούμε από μια προσέγγιση βάση έκθεσης ανάγκης από το θεσμικό όργανο αυτό για το μέλλον του περιοδίστου συνομικού πλαισίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν στην πρόσφατη πρόσφαση της για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και η ομάδα υψηλόβαθμων αξιωματούχων αναγνωρίζουν ότι οι διαδικασίε και διατάξει για την παροχή και όλα τα κρατη ωφελούνται από τη δράση των κρατών μελών που υποστηρίζονται από τον εθνικό προπολογισμό. Γιατί είτε δεν τα, τα εξωτερικά σύνορα, είτε υλοποιούν το κεκτημένο για το άσυλο. Ε, κάνουν δηλαδή και διεκπεραιώνουν αιτήσει άσυλο, αναγνωρίζουν ε, σε μεγάλο βαθμό, σε υπερβολικό βαθμό, σε παροχές και ποσά έκτακτης ανάγκης. Αυξήθηκαν λοιπόν τα απόστημά τους, χρησιμοποιήθηκαν αυτές τις ενισχύσει έκτακτης ανάγκης και μία επισκόπηση όλων των ε, προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν μεταξύ 2014 και 2016 για το ΆΜΙΦ και το ISF αποκαλύπτουν ότι πέρα από την Ελλάδα και την Ιταλία και η Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, έχει ενίσχυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ε, λειτουργική κατάρτιση της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης. Ε, αυτό είναι γενικό φαινόμενο, δεν εστιάζεται μόνο σε κάποια κρατημέλη. Αυτές οι μεγαλύτερες ανάγκες λοιπόν δεν είναι μια έκτακτη ανάγκη. Θα συνεχίσουν να ε, παρουσιάζονται, θα γίνουν αυξημένη ενίσχυση μέσω των υπηρεσιών αυτών. Και αυτό συνδέεται και με την ειδική αυτή ενίσχυση, την ενίσχυση έκτακτης ανάγκης. Αυτές οι ενισχύσεις ακόμα αποκαλούνται έκτακτης ανάγκης, παρά το γεγονός ότι κάποια κρατημέλη όπως η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν μόνο προσωρινές είναι αυτές οι υπηρεσίες. Χρησιμοποιήθηκαν και, άλλα, και άλλοι δύο-δύο, όπως ο μηχανισμός ε, ε, αστικής προστασίας, προστασίας του πολίτη ε, που φυσικά έχει τα όρια του, γιατί χρησιμοποιεί μόνο μη οικονομικής ε, πόρους, όπως για παράδειγμα εξοπλισμός, προστασία του πολίτη, ε, που φυσικά έχει τα όρια του, γιατί χρησιμοποιεί μόνο μη οικονομικής πόρους, όπως για παράδειγμα εξοπλισμός και εξαρτάται φυσικά και από την εθελούσια συμμετοχή και συνεισφορά των κρατών μελών. Η ανταπόκριση λοιπόν στις ανάγκες αυτές ήταν σε διάφορες περιπτώσεις ανεπαρκής. Πιστική βοήθεια και υλοποιήθηκαν παρά αυτά κατά την εισρωή μεταναστών και προσφύγων, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα έκτακτο εργαλείο με περίοδο δραστηριοποίησης ε, τριών ετών. Το 2019 θα τερματιστεί μέχρι τον Απρίλιο 2000. Αρρωγή σε τρόφιμα, μη τροφική αρρωγή, καταλήμματα και υποστηρίχθηκε από διάφορες ενώσεις μεταξύ των οποίων υπό εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο και αυτό μπορούμε να το δούμε και από άλλες γραμμές του προπολογισμού και από άλλα ταμεία, από τα τραφετικά ταμεία τι έχει συμβεί αντίστοιχα υπό εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο και αυτό μπορούμε να το δούμε και από άλλες γραμμές του προπολογισμού και από άλλα ταμεία, από τα τραφετικά ταμεία τι έχει συμβεί αντίστοιχα. Επίσης, δίκαιη κατανομή μέσω απλούστευση τη διαχείριση των ε, ταμείων και των πόρων, το συστήματα ελέγχου και διαχείρισης τα οποία εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη και πρέπει να εφαρμόσουν είναι πάρα πολύ περίπλοκα και προαπαιτούν μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό για να λειτουργήσουν. Από, υπό την έννοια λοιπόν αυτή κοστίζει χρήματα να απορροφηθούν ε, οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εναρμόνιση των διάφορων ε, γραμμών του προπολογισμού, όπω προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι ένα βήμα προ σωστή κατεύθυνση. Φυσικά μέσα στην εναρμόνιση αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί η λιγότερο ε, περίπλοκη διαδικασία. Τέλο, συμπληρωματικότητα με τι εθνικέ χρηματοδοτήσει σε ό,τι αφορά και τα τι εξωτερικέ υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είπε και ο διευθυντή τη Frontex. Πολύ σημαντικό στοιχείο και συμπληρωματικότητα μεταξύ των εργαλείων, όπως είναι για παράδειγμα και με τα άλλα ταμεία, όπως τα τα ταμεία. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να δημιουργούν συνέργειες. Σκοπός μας είναι να περάσουμε από τις συνέργειες και από εξάρτηση σε πόρους έκτακτης ανάγκης, όπως το εργαλείο έκτακτης ανάγκης, σε πλήρη συμπληρωματικότητα με μόνιμους γραμμές του προπολογισμού, όπως είναι αυτές στο πλαίσιο στις ε, πολιτικές συνοχή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ τους ε, πέντε μιλητέ μας που μας μίλησαν για τις εμπειρίες τους. Εδώ ψηφίζουμε τις πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου, αλλά αυτοί μας λένε πώς ε, τις ξοδεύουμε. Τώρα, θα ξεκινήσει η συζήτηση. Ιταλίας-Γαλλίας, κοντά στη Βεντιμίλια. Και εκεί μαζί με τον Ιταλό συνάδελφο, τον κύριο Βιώτη, συναντηθήκαμε με Γάλλους και Ιταλούς ε, εκεί εκπροσώπους. Ε, προσπαθούμε να βάλουμε στην αστυνομική βάση ε, μία γραμμή, ούτως ώστε να εμπλακούν περισσότερο οι τοπικές αρχές. Θα δούμε σε ποιο βαθμό οι συμφωνίες του Δοβουλίνου για τα σύνορα γίνονται σεβαστές. Ε, έχουμε σύνορα μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας, ότι τους διακινητές. Εδώ έχουμε το Γενικό Διευθυντή της ε, Frontex. Όταν έχετε όταν στέλνετε κόσμο στα εξωτερικά σύνορα, δικούς σας ανθρώπους, ε, φοράνε τη στολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ορατή στα εξωτερικά σύνορα. Κύριε Λετζέρη, προσπαθούμε να δείξουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι ορατή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αξιωματικοί που πηγαίνουν στι επιχειρήσεις τη Frontex, έχουν και ένα γυλαίκο στη διάθεσή τους, έχουν και ένα κοιτίο με το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τα πλοία, που είναι αυτό που κοστίζει περισσότερο έτσι, από τον τεχνικό εξοπλισμό. Είχαμε κάποιες ε, τεχνικές αλλά και νομικές δυσκολίες. Μερικές φορές αναγκάζομαι να πιέσω λίγο τα κράτη-μέλη να κάνουν κάποια πράγματα. Κάποια από τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη με ρωτάνε τι σημαία να βάλουμε σε αυτά τα σκάφη. Ε, είναι πάντως έτοιμα να βάλουν την ε, σημαία της Ευρώπης. Σίγουρα θα πρέπει η Ευρώπη να φαίνεται, ε, ειδικά σε αυτές τις δράσεις που γίνονται υπό την αιγίδα της Ευρώπης. Κύριε ευχαριστώ πολύ. Να μου επιτρέψετε να συνεχίσω στα τσεχικά, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, όπως σας εξήγησα να μιλήσω τσεχικά, ήθελα και με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Αθηναίων που ε, βρέθηκε κοντά μας. Πριν από τρεις εβδομάδες πέρασα από την Αθήνα. Πήγα και στη Δέσβο στα δύο hot spot και θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στα πρόσωπα τα οποία φροντίζουν τους ε, πρόσφυγες στα μέρη αυτά. Πήγα στην Αθήνα στον Ελαιώνα. Πήγα και στην βάση του Frontex. Η ερώτησή μου προς τον εκπρόσωπο του Frontex έχει ως εξής. Ξέρουμε ότι επεκτείνεται, δηλαδή επεκτείνει τον αριθμό ε, προσώπων που απασχολεί ο Frontex. Ρωτώ λοιπόν, το προσωπικό του Frontex στο μέλλον θα είναι γραφειοκράτες ή θα είναι αστυνομικοί και συνοριοφύλακες. Θα είναι διοικητικοί υπάλληλοι ή θα είναι επιχειρησιακοί, δηλαδή θα βρίσκονται πραγματικά στα σύνορα. Εν τέλει, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλη μεταναστευτική πίεση που προέρχεται από την Τουρκία. Ιδίως τα ελληνικά νησιά αλλά βέβαια και τα χερσαία σύνορα της Ελλάδος αντιμετωπίζουν αυτήν την πίεση. Χερσαία σύνορα τα οποία δεν φυλάσσονται επαρκώς. Πράγματι, τα μεταναστευτικά ρεύματα έχουν αυξηθεί τόσο που πλέον τα hot spot δεν είναι ικανά να υποδεχθούν τους αριθμούς αυτούς ανθρώπων. Άρα με αυξάνει και η πίεση επί των συνοροφυλάκων και ακτοφυλάκων. Σας ευχαριστώ πάντως για το έργο που κάνετε. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ορατή με τον τρόπο αυτό. Οι δε άνθρωποι που συνάντησα στην επίσκεψή μου αυτή είναι γνώμονες για την χρηματοδοτική υποστήριξη. Αυτόν που επικρίνουν είναι η ελληνική κυβέρνηση λόγω της κολυσιεργίας της. Ευχαριστώ κυρία Βεργιά. Κυρία Πρόεδρε, βλέπω ότι και ο πρόεδρος Αρτουή απεχώρησε. Θα ήθελα να του πω όμως ότι αν αποκατασταθούν τα εσωτερικά ο κύριος Αρτουή, δεύτερο σχόλιο. Όντως υπάρχει πρόβλημα ορατότητας των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Το ζήτημα που θέτω εγώ είναι ότι στη μεγάλη δίνονται, χορηγούνται στις χώρες μέλη που μετά κατανέμουν τα κονδύλια αυτά κατά βούληση. Τέλος πάντων όχι ακριβώς κατά βούληση, αλλά χωρί να λένε απαραίτητα ότι πρόκειται για ευρωπαϊκά χρήματα. Έχω πάει κατά επανάληψη στο Καλέ και έχω συναντηθεί και με την νομάρχη του Καλέ και μάλιστα και μέσα σε μια αποστολή της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών με ρώτησε λοιπόν η Νομάρχη γιατί δεν βοηθάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φέρα προβλήματα και σε ό,τι αφορά την κατανομή και σε ό,τι αφορά τι αιτήσει. Ε, θα ήθελα να τα δούμε λιγάκι αυτά τα θέματα μαζί με τον κύριο Λετζέρι από τη Frontex. Αυτή τη στιγμή κοιτάμε τις κατανομές της Κομισιόν. Τα σχέδια τέλο πάντων, το σχεδιασμό τη Κομισιόν. Υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στις πιστώσεις ε, στον επόμενο πολυετή, στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε 10... Ο, δηλαδή, το, ζητήσατε αυτό. Το ζητήσατε αυτό το νούμερο ή απλώς ένα στρογγυλό νούμερο, ας πούμε. Με ποια κριτήρια 10, θέλετε 10.000 άτομα, ας πούμε, να έχετε. Επίσης, εάν αυτό προβλέπετε, Πώ θα εξασφαλίσει και, όταν, και θα τα έχουμε κατανοεί με βάση τα σημερινά προβλήματα τη σημερινή κρίση. Και όταν θα ε, εμφανιστεί η επόμενη κρίση, θα είναι αλλού, α πούμε. Και δεν θα είναι απόλυτα χρήσιμα αυτά τα άτομα. Γιατί δεν θα έχουμε την κατάλληλη ευελιξία να μετακινούμε άτομα στην κατάλληλη ε, το πλαίσιο. Κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Προ τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε, κύριε Χάουαρτ. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Μία στην πραγματικότητα. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες για την απορρόφηση των κονδυλίων, για την εφαρμογή των κονδυλίων. Γιατί δεν έχει η Κομισιόν ένα κατάλληλο μηχανισμό για την υποβολή εκθέσεων, ούτω ώστε να μπορούν οι συνομοθέτε να παίρνουν σωστέ αποφάσεις για τα θέματα του προπολογισμού. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Έχουμε τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και τον εκπρόσωπο της Frontex. Θα θέλανε αυτοί οι δύο κύριοι να μας απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις που ακούσαμε. Καταρχάς ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Μήπως μπορεί να απαντήσει. Κυρία. Δηλαδή. Σας ευχαριστώ και να απαντήσουμε σιγά σιγά τις ερωτήσεις της κυρίας Γκρέσλε. Να ξεκινήσω καταρχάς ε, και να μιλήσω για την δυνατότητα που έχουν και οι Δήμοι να λάβουν χρήματα από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Αυτό επιτρέπεται μέσω του ΑΜΕΦ, αλλά πάντα υπό τον έλεγχο των εθνικών αρχών. Υπάρχουν ε, χώρες όπου οι εθνικές αρμόδιες ε, οι υπηρεσίε οι οποίε διαχειρίζονται τα ταμεία ΑΜΕΙ συνεργάζονται με Δήμου και κοινότητε για τη διάθεση πόρων. Άλλε το κάνουν λιγότερο αυτό, αλλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα και υπάρχει προφανώ και. Ε, αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί και την επόμενη διαμορφώση των ταμείων. Είναι προφανέ ότι αυτό χρειάζεται. Φυσικά ανακύπτει και το θέμα του ποιο ελέγχει τελικά τη ροή των πόρων, γιατί μετά περιορισμένους πόρους που έχουμε δεν μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε όλα. Σε ό,τι αφορά την υπατερμοστία του ΟΕΕ. Έχουν παρουσία και στα νησιά. Δεν μπορώ να σας αναφέρω όλες τις λεπτομέρειες όλων των συμβάσεων που έχουμε, αλλά η υπατερμοστία έχει μεταβεί εκεί για να αυξήσει την δυνατότητα υποδοχή. Το μεγαλύτερη σύμβαση που έχουμε είναι για την υπηρετική Ελλάδα, όχι για τα νησιά, όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη για προσφυγικούς καταβλισμούς για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που καταστάνουν στην υπηρετική Ελλάδα. Η κατανομή των μέσων, η κλίδα ορίστηκε, ορίστηκε στην νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2013. Έχουμε τα άτομα τα οποία αιτούνται άσυλο, τα άτομα τα οποία πρέπει να ενταχθούν, τα άτομα τα οποία επιστρέφονται. Άρα εξαρτάται το θέμα. Το πρόβλημα είναι η περίοδος ε, η οποία επιλέχθηκε, γιατί αυτό έχει να κάνει πάντα με τη στατιστική περίοδο 2010-2011. Προφανώ τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ από τότε και αυτό είναι ένα σημαντικό μάθημα το οποίο ε, αποκομίζουμε για την επόμενη πρόταση, την επόμενη νομοθετική πρόταση για την Ταμεία από πλευρά του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η περίοδος που χρησιμοποιείται ως βάση για την κλειδά κατανομής για την εκχώρηση των πόρων θα πρέπει να είναι ευέλικτη, θα πρέπει να είναι προσαρμόσιμη ανάλογα και με τις εξελίξεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, πιστεύουμε ότι θα χρειαστεί ένας τεχνικός, ε, ε, μια τεχνική προσαρμογή, γιατί προφανώς μα απασχολεί ιδιαίτερα και έχει ασκηθεί και μεγάλη κριτική κατά του γεγονότος αυτού. σε ό,τι αφορά την, ε, ε, ε, ε μας, την αρρωγή εκτίθεση Προφανώς μας απασχολεί αυτό και προφανώς έχουν καεί κάποια προγράμματα, έχουν εξευρεθεί 100% και Άρα η αρρωγή αυτή της ανάγκης δεν είναι μέτρο έκθεση ανάγκη, αλλά συμπληρωματικό μέσο για να εξασφαλίσουμε ότι τα επιπλέον καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη μπορούν να συγχρηματοποτηθούν. Αλλά γενικά ο στόχος μας, το είπα και προηγουμένως, είναι να περάσουμε σε ένα καθεστώς μιας στρατιωτικής βοήθειας και διαμορφωσής ε, της κατάστασης. Το ερώτημα της, το ζήτημα της διαφάνειας. Άκουσα τι είπατε. Προφανώς θα πρέπει να εργαστούμε καλύτερα. Δεν είναι εύκολο να παραμένουμε πάντα ενήμεροι σε ό,τι αφορά και την κατάσταση που μεταβάλλεται στα κράτη-μέλη αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί πάντα να ε, καθορίζει πόσο τελικά έχουμε δώσει στα κράτη-μέλη κάθε χρόνο. Αυτή η απόφαση λαμβάνεται τέλη Μαΐου, αρχίες Ιουνίου ε, κάθε φορά και χορηγούνται τα ανάλογα ποσά στα κράτη-μέλη. Αλλά όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές είναι μεγάλο και δύσκολο έργο αυτό. Ευχαριστώ. Περικά σύνορα. Αυτό που κάναμε τώρα με το επιπλέον προσωπικό είναι ότι δώσαμε περισσότερο κλασικό μοντέλο δηλαδή, που έχουμε, το, το ότι χρησιμοποιούμε δηλαδή συνοριοφύλακες από τα κράτη-μέλη, έχει φέρει στα όρια του ε, το δυναμικό αυτό το πόστο μου. Τον Ιανουάριο του 2015 θυμάμαι ότι μπορούσαμε να στείλουμε περίπου 350 αξιωματικούς. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό το εξήγησαν και άλλοι παρόντες εδώ, ε, ομιλητές. Πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει με αυτή την έννοια, με αυτό το... μια κεντρική μονάδα την αιτία να την υποδεχτεί και να τη φιλοξενήσει το, η Frontex. Είναι τμήμα των, της διαχείρισης λοιπόν είναι τεμπέληδες ή τα πίνουν, ας πούμε, σας ε, καθησυχάζω όλους. Μόνο τέσσερις αξιωματικοί. Ε, δεν επιλέγουμε τέτοιου ανθρώπου. δεν θέλουμε τέτοιου ανθρώπους. Πρέπει να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, αντιμετωπίζουμε και τέτοια προβλήματα. Όταν έχεις, ας πούμε, 1.500 ανθρώπους, ε, δεν ξέρει όταν υπάρχουν τέτοιου τύπου προβλήματα. Ευχαριστώ. για την πολύ ενδιαφέρουσα πρόσθετη παρέμβασή σας. Θα αρχίσουμε τώρα το δεύτερο πάνελ λέει η κυρία Κούντρισκα, αλλά παραδίδει το μικρόφωνο στην κυρία Γκρέσλε. Θα προχωρήσουμε τώρα στη συζήτηση ε, περί κονδυλίων. Χαίρομαι που είναι παρούσα η κυρία Λαμάρκ, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχει συντάξει και σχετική έκθεση. Παρακαλώ ωστόσο να μην υπερβεί το όριο των 10 λεπτών. Euh, Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην μεταναστευτική κρίση ε, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει κατεπίγουσες ε, καταστάσεις και προβλήματα τρομακτικής ε, δυσκολίας και εμβέλειας. πολλαπλασίασε τα ποσά σε διάφορους τομείς και τις, τους οργανισμούς, νέα χρηματοδοτικά μέσα, ε, στοχευμένες δράσεις για τα hot spot και μια προσπάθεια κινητοποίησης των ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων. Το ελεκτικό συνέδριο, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία αυτών των θεμάτων, έβαλε το θέμα της μετανάστευσης και του ασύλου στις προτεραιότητες ε, ελέγχου. Και από το 2016 ε, ξεκινήσαμε καμιά δεκαριά εργασίες για τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου και συναφή θέματα όπως παραδείγματο χάρη την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης. Στην ετήσια έκθεση για την, ε, το 2016, πέρυσι, για πρώτη φορά βάλαμε ένα κεφάλαιο για το MFF3, δηλαδή ασφάλεια και ηθαγένεια. Θα κάνουμε το ίδιο και φέτος. Ε, βγάλαμε πολλές εκθέσεις το 2017 και μια ειδική έκθεση για τα hot spot, τα, κυρίως τα σημεία υποδοχή στην ε, ε, Ελλάδα και στην Ιταλία. Έχουμε τρει ειδικέ εκθέσει. Ένα για την, ε, το μηχανισμό υπέρ των προσφύγων στην Τουρκία, για το καταπίστευμα τη Αφρική που θα βγει στο τέλο του 2018 και επίση, επειδή μα το ζήτησε η, Κομισιόν, η Επιτροπή μάλλον Λίμπε, μία έκθεση για τα, τα συστήματα πληροφόρηση που χρησιμοποιούμε στα εξωτερικά σύνορα που θα δημοσιευθεί τον Απρίλιο. Ε, αύριο θα ετοιμάσουμε ενημερωτικό έγγραφο για την ένταξη των μεταναστών που μελετά τη χρήση του Ταμείου ΑΜΙΦ, το οποίο συζητήσατε σήμερα, και επίση κάθε χρόνο ετοιμάζουμε εκθέσει για του οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι τα συμπεράσματα από όλε αυτές τις εργασίε ε, στην ειδική έκθεση για τα hot spot Είδαμε τη θετική επίπτωση που είχε αυτή η επιχείρηση στην Ιταλία και στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις και κάποιες αδυναμίες σε ό,τι αφορά ιδίω τους ασυνόδευτους ανήλικους. Τα σημεία αυτά, τα hot spot, δηλαδή συνεισέφεραν στο να ε, βελτιωθεί η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ιταλία και στην Ελλάδα που είναι στην ε, πρώτη γραμμή του πυρός ε, μπόρεσαν να αυξήσουν το, τη δυνατότητα υποδοχής, να βελτιώσουν τις διαδικασίες καταχώρησης και βελτίωσης του συντονισμού της βοήθειας. παρόλα αυτά χρειάζονται περισσότερα μέσα γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Το ελεγκτικό συνέδριο συστήνει λοιπόν στην Ελλάδα να αυξήσει το δυναμικό υποδοχής της, να βελτιώσει τις υποδοχές ε, στέγασης, να μειώσει τις ε, προθεσμίες ε, επεξεργασίας των αιτήσεων με τη βοήθεια της ΕΑΣΟ, να ενημερώσει καλύτερα τους ετούντες, στην Ιταλία να αυξήσει τα σημεία εισχώρησης. Επίσης, ε, να βελτιώσει την ε, υποδοχή των ασυνόδευτων ε, ανηλίκων, να έχουν περισσότερους εμπειροχνόμενους στα κράτη-μέλη και επίσης να αξιολογήσει όλο το μηχανισμό και να βγάλει διδάγματα. Δεύτερη παρατήρηση για όλες τις εργασίες μας. Από όλες τις εργασίες μας βλέπουμε εδώ και καιρό την περιπλοκότητα της χρηματοδότησης και τη δυσκολία να εντοπίσουμε τις δαπάνες που αφορούν τις συγκεκριμένες δράσεις. Λόγω του ότι έχουμε πάρα πολλά ταμεία τα οποία χρησιμοποιούνται πέρα από το ΑΜΙΦ και το κοινωνικό ταμείο. Γιατί μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ταμείο της ένταξης, ε, ανάπτυξης, ε, το ΦΕΝΤΕΡ, το Έρασμους, την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και άλλα και άλλα. Φερρυπίν, στην έκθεσή μα για τον προπολογισμό του 2016 διαπιστώνουμε ότι η Κομισιόν δεν μα είπε το συνολικό ποσό των ταμείων που κινητοποιήθηκε για να καλύψουμε την κρίση, τον, την προσφυγική και την μεταναστευτική του 2016 και εσωτερικά και εξωτερικά και είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε μια αξιολόγηση, μια εκτίμηση ας πούμε του ποσού αυτού. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει μια ειδική δομή για να διαβιβάζονται αυτές οι πληροφορίες ούτως ώστε να συνειδητοποιούμε πώς χρησιμοποιούνται τα ταμεία. Και να χρησιμοποιούμε τον ΩΣΑ, τα στοιχεία του ΩΣΑ, ε, μόνο για θέματα μετανάστευση και απασχόληση. Ε, γιατί δεν είναι κατάλογοι όλα τα θέματα. Επίση, ε, οι μηχανισμοί χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ περίπλοκοι. Είναι ένα σύνολο μηχανισμών που συνδέεται με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό ε, αλλά έχει και δικά του στοιχεία. Αυτό το λέμε ξανά και το λέει και η Επιτροπή Προπολογισμών και είναι ένα μηχανισμό που περιορίζει τη διαφάνεια και τον έλεγχο. Ακριβώ γι' αυτό. Συχνά γνωρίζουμε μόνο τις πληρωμές που αφορούν τα βασικά ταμεία, δηλαδή το ταμείο ας πούμε αμύθ, αλλά δεν γνωρίζουμε τη χρηματοδότηση ε, από άλλες πηγές που προέρχονται συχνά από άλλους τομείς. Επίσης για το αμύθ στα κράτη-μέλη δεν μπορούμε να διακρίνουμε τις προκαταβολές από τις ε, τελικές πληρωμές, γιατί δεν αποσυνδέουμε τα, τις μένα από τις δε. Επίσης, ε, έχουμε πρακτικές διαχείρισης προβληματικές στους διάφορους οργανισμούς. Η Frontex, ε, με βάση τις παρατηρήσεις που κάνουμε για τη χρήση των επιχορηγήσεων, το 2015 ξεκίνησε μια διαδικασία διαγωνισμών ε, θα πρέπει, κάνει δηλαδή διαγωνισμούς ούτως ώστε να ε, προσλαμβάνει ας πούμε να έχει υπηρεσίες α, καλύτερες. Παραδείγματο χάρη να έχουμε λιγότερα μεγάλα σκάφη ας πούμε. Ε, όχι τόσο μεγάλα όπως αυτά που δίνουν τα κράτη-μέλη ας πούμε. Θα πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση εκπόστε ε, για όλα αυτά εκ των υστέρων αξιολόγηση δηλαδή για τη Frontex και για τα hot spot και να γίνει επίσης και αξιολόγηση ε, σωστή των κρατών, μελών. Γιατί έχουμε διαφορετικούς δείχτες από κράτος σε κράτος. Ε, επίσης, ανταλλάσσουν δεδομένα η Frontex και τα κράτη-μέλη για την ε, καταχώρηση των λαθρομεταναστών. Ε, συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι συνολικά η Ένωση μπόρεσε να προσαρμοστεί στην ε, κρίση και στην, ε, στην κατεπίγουσα ανάγκη και να διευκολύνει την υποδοχή των ε, μεταναστών, αλλά υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις και δεν μπορέσαμε ούτε ποσοτικά ούτε ποιοτικά να ανταποκριθούμε σε όλες τις ανάγκες. Οι διαδικασίες είναι πολύ προβληματικές, καθυστερούν, δεν πλαισιώνουμε σωστά τους ασυνόδευτους ανήλικους και χρειάζεται επιπλέον προσπάθεια και από την Ένωση και από τα κράτη-μέλη. Είναι σαφές ότι η ευελιξία στη χρήση των ταμείων είναι καλή για να αντιμετωπίσουμε τις κατεπίγουσες ανάγκες, όμως αυτή η ευελιξία γίνεται εις βάρος μια σωστής ε, και έφτακτης διαχείρισης ε, και αυτό δεν γίνεται γιατί υπάρχει φοβερή περιπλοκότητα, αδιαφάνεια, υπάρχουν πάρα πολλά ταμεία τα οποία κινητοποιούμε και που δεν έχουν πάντα άμεση σχέση με τη συγκεκριμένη δράση που προωθούμε και τέλος έχουμε δυσκολίες να συνειδητοποιήσουμε τη χρήση των πιστώσεων και των ε, δαπανών και αυτό ε, δυσκολεύει τον έλεγχο και περιορίζει την πληροφόρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμπερασματικά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα εξορθολογισμό Μία προσπάθεια διαφάνειας και σωστής αξιολόγησης. Αυτό είναι απαραίτητο για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των μεταναστευτικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενημέρωση των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λαμάρκ. Ηνωμένων Εθνών για του πρόσφυγε, Έχετε το λόγο. Okay, sorry. Yes. Um, yes, good afternoon. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Εκπροσωπώ το γραφείο του ΥΠΑ του Αρμοστή των ε, Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μας απευθύνατε. Ο ΥΠΑΤΟΣ Αρμοστής είναι διεθνής παρατηρητής του μηχανισμού χρηματοδότησης. Άμεσα ενδιαφερόμενο μέρος και δικιούχος. Είτε πρόκειται για emergency funding, είτε για κοινή χρηματοδότηση και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν σχετική εμπειρία. Θα προσπαθήσω να φωτίσω ορισμένες πτυχές του θέματος. Κάποια τα είπατε ήδη. Ορισμένα θα πω ακόμη για να ε, ξεκαθαρίσω περισσότερο ποια είναι τα ζητήματα της αποτελεσματικότητας. Ε, ποιες είναι οι αρχές για τη χρήση των χρημάτων. Θα αρχίσω από εκεί που τα άφησε η προηγούμενη συνάδελφός μου. Μίλησε δηλαδή για την αρχή της προστιθέμενης αξίας και της προσθετικότητας των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Είναι σημαντικές έννοιες αυτές ε, σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Έχουν συζητηθεί βέβαια και από πολλά χρόνια ήδη και θα συνεχίσουν να συζητούνται και για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όμως για μετανάστευση και άσυλο έχουν και εκεί τη σημασία τους και πρέπει να διευκρινιστούν. Τα λέγω αυτά διότι στα πλαίσια της ε, κοινή διαχείρισης τα χρήματα αυτά φέρονται συχνά ως ότι δίθεν απορροφώνται και εξαφανίζονται μέσα στους εθνικούς προϋπολογισμούς, ενώ δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν τα ευρωπαϊκά χρήματα τα εθνικά, ούτε να τα συμπληρώνουν. Τους εθνικούς προϋπολογισμούς για άσυλο και μετανάστευση. Αυτά εισαγωγικά. Επιθυμώ να πω επίσης ότι αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα δεν μπορούν να στερούνται ωστόσο νομιμότητας. Ενώ δηλαδή ότι η νομιμότητα της χρήσης των ευρωπαϊκών χρημάτων και για ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να είναι στην βάση πάντοτε των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να συμμορφούνται με τις σχετικές διατάξεις και για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα εφόσον επιλέξουμε μια ολιστική προσέγγιση. Επιτρέψτε μου να γίνω πιο συγκεκριμένη σχετικά με το Ταμείο ΑΜΙΦ. Ορισμένοι μίλησαν για την ανάγκη καλύτερου προγραμματισμού, για χρήση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων μέσα στον δημοσιονομικό κύκλο. Αυτό είναι σημαντικό, να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές. Έχω και μία σύσταση προς τις ίδιες τις χώρες μέλη, που δεν έχει γίνει ακόμη, ότι δηλαδή οι χώρες μέλη, στο βαθμό του δυνατού, θα πρέπει να αναθέτουν την διαχείριση των χρημάτων σε εμπειρογνώμονες. Ας μην αφήνουν τα πράγματα αυτά μόνο στα χέρια του Υπουργείου Οικονομικών, κάτι που γίνεται συχνά με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Εδώ είναι πολύ σημαντικό όμως να πάνε τα χρήματα σε αυτούς που γνωρίζουν που θα πρέπει να διαθέσουν τα κονδύλια και τι θα τα κάνουν. Κάτι το οποίο θα επιτρέψει και την συντόμευση των διαδικασιών, την ε, απάλληψη δηλαδή των καθυστερήσεων. Συχνά οι καθυστερήσεις, λέγουν ορισμένοι, είναι αναπόφευκτες. Όμως ε, ε, επιφέρει μεγάλη ζημιά σε αυτούς οι οποίοι εργάζονται ε, επιτόπου στο πεδίο. Ορισμένες μη κρατικές οργανώσεις και τοπικές οργανώσεις αντιμετώπισαν σοβαρότητα προβλήματα λόγω των καθυστερήσεων αυτών. Τονίζω επίσης κάτι το οποίο λέχθηκε ήδη, αλλά εννοώ ανάγκη περισσότερης ενημέρωσης, διαφάνειας και ίχνηλασιμότητας. Δηλαδή γνωρίζουμε, αλλά δεν πρέπει να γνωρίζουμε για το που χρησιμοποιούνται τα χρήματα, αλλά πρέπει να μπορούμε να συναγάγουμε και τα σχετικά συμπεράσματα. Σε 1,5 χρόνο, το 2019, θα έχουμε ακόμα Δηλαδή, τέλο πάντων, έχουμε ακόμα μέχρι το 2020 2,5 χρόνια και ακόμα δεν έχουμε την ενδιάμεση έκθεση η οποία θα εκδοθεί κάποια στιγμή του επόμενου μήνε. Δεν έχουμε πληροφορίες ούτε για τους μηχανισμούς παρακολούθησης, ούτε για την αξιολόγηση που γίνεται της ε, δαπάνησης των χρημάτων που γίνεται από τις διαχειριστικές αρχές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να πω ακόμη κάτι που είναι πολύ σημαντικό για το ΑΜΥΦ και έχει σχέση και με το Ταμείο Συνοχής και πρόκειται για την αρχή της συνεργασίας, partnership principle. Αυτό μάλιστα περιλαμβάνεται και στην νομική βάση του ΑΜΙΦ υποτίθεται ότι είναι ένας συμβουλευτικό μηχανισμός στον οποίο συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή και οι φορείς της ε, κοινωνία των πολιτών, οι τοπικές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι και οι κοινωνικοί φορείς. Αυτό όμως ο συμβουλευτικό ε, μηχανισμό πρέπει να γίνει δεσμευτικό, όπω γίνεται και το Ταμείο Συνοχή, διότι θα αποτελέσει ένα μηχανισμό που θα παρακολουθεί την χρήση των χρημάτων και, επομένως, ε, και ε, ενδεχομένως θα επιφέρει και διορθώσεις. Αυτό θα βελτιώσει την αποδοτικότητα χρήσης των χρημάτων. Ήδη αυτά περιλαμβάνονται στο ΑΜΥΦ. Όμως εφαρμόζεται σε τελείως διαφορετικά επίπεδα. Σε ορισμένες χώρες μέλη έχει γίνει κάποια ενημερωτική συνάντηση και αυτή η ενημερωτική συνάντηση θεωρήθηκε ότι ικανοποιεί την πρόβλεψη του νόμου για τον συμβουλευτικό μηχανισμό, που δεν αρκεί όμως. Θα ήθελα επίσης να τονίσω την ανάγκη περιορισμού της γραφειοκρατίας. Μεταφέρομαι το μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έντονα ότι χρειάζονται ειδικέ δεξιότητες για την διαχείριση των ευρωπαϊκών χρημάτων και για να μπορεί να γίνει αυτό βεβαίως πρέπει να γίνει σχετική εκπαίδευση των στελεχών. Άρα, για να χρησιμοποιήσει κανεί ευρωπαϊκά χρήματα, πρέπει να δαπανίσει πρώτα χρήματα για την εκπαίδευση, ξαναλέω. Για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα, θα πρέπει να υπάρχει και ένα ελάχιστο ποσοστό χρημάτων σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών και σε τοπικούς φορείς. Αυτό έχει ξαναλεχθεί, έχει λεχθεί κατ' επανάληψη. Αν δεν υπάρχει όμως ένα ελάχιστο μερίδιο, εκεί βέβαια με κάποια ευκαμψία, αλλά αυτοί που βρίσκονται στην πρωτοπορία της προσπάθειας πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα αναγκαία εργαλεία και βεβαίως και να μπορούν και να δικαιολογήσουν απέναντι στους πολίτες για ποιο λόγο έχουν το, τη δυνατότητα αυτή. Τέλος, η Γενική Διεύθυνση Home, η χρηματοδότηση του ΑΜΥΦ και η εξωτερική διάσταση, δηλαδή η δραστηριοποίησή του εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει και αυτά να έχουν ένα συντονισμό. Τελειώνω με δύο θέματα, διότι εδώ εξετάζουμε το επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή όχι μόνο το αμύφ ή μάλλον να το πω καλύτερα αμφ, διότι η λέξη integration φεύγει, επομένως αυτό το γιώτα του integration φεύγει και πηγαίνει στο Ταμείο Συνοχής. Εδώ έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις. Είδαμε στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το Ταμείο Συνοχής θα μειωθεί το λιγότερο κατά 7% λόγω Βρετανικής αποχώρησης. Πώς λοιπόν θα κάνουν όμως περισσότερα πράγματα με λιγότερα χρήματα και όταν λέω περισσότερα διότι θα μπει εκεί το integration, αυτό το I που θα φύγει από το AMIF. Αυτή λοιπόν είναι μια ερώτηση προς αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις αλλά μπορεί και να αποδυναμωθεί και να λησμονηθεί στα πλαίσια του ΑΜΥΦ προβλέπεται 20% υποχρεωτικών δαπανών για και αποδοτικότητα των δαπανών στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος Γκρέσλε. Το παρουσιάσατε με πάρα πολύ ταχύς ρυθμούς, αλλά ευτυχώς τα να παραδειρμενείς. Να δώσουμε το... Που μας προσκαλέσατε. Εκπροσωπώ την ΣΕΠΣ που είναι ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψεως. Είμαι ερευνήτρια για σχετικά θέματα στην ΣΕΠΣ. Έχουμε κάνει ορισμένες μελέτες και ορισμένες από αυτές για τις εξωτερικές πτυχές της ε, χρηματοδότησης θεμάτων μετανάστευσης και έγιναν θετικά δεκτές και από την Επιτροπή σας των Προϋπολογισμών και από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και όταν προσκληθήκαμε σήμερα να συζητήσουμε θέματα εσωτερικά της χρηματοδότησης των θεμάτων μετανάστευσης, αναζητήσαμε τι ήταν αυτό που διέπει τις ε, μελέτες μας έως τώρα για θέματα κράτους δικαίου, για νόμιμη μετανάστευση, για διαχείριση ε, του χώρου Σένγκεν και άλλα σχετικά και θα θέλαμε να εξαγάγουμε ορισμένα συμπεράσματα διαπιστώσαμε ότι ένα από τα πιο βασικά είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτιμοποίησης αυτής της χρηματοδότησης. Που είναι περίπλοκη υπόθεση. Όπως λοιπόν έλεγα και όπως τονίζεται συνήθως, κύριε του κράτους δικαίου και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνεδρίο αλλά και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής το τονίζουν αυτό ότι για την βελτίωση της νομοθεσίας η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα σημαίνει και τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτά τότε χρηματοδότηση ανεξάρτητων οργανισμών αλλά με την διατήρηση των ίδιων των προτύπων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως του κώδικα των συνόρων Σέγγεν κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου κλπ. Διδάγματα από την ε, λειτουργία μας επιτόπου. Εμείς ε, κάναμε άλλη μία μελέτη που επιγράφεται Anti-Smuggling Policies και βλέπετε το γράφημα ε, σχετικά ασφαλείς σχετικά με το ότι κάνουν. Ένα από τα διδάγματα λοιπόν είναι ότι η χρηματοδότηση της μετανάστευσης έχει σχεδιαστεί υπό την υπόθεση ότι οι χώρες μέλη σέβονται την νομιμότητα και την ανεξάρτησία των ε, ε, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, όπως η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ασύλου και ενσωμάτωση των προσώπων αυτών. προτεραιότητα της ασφάλειας είναι σημαντική. Αλλά ασφάλεια για ποιον. Διότι βλέπουμε ότι οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών αυτών που προσφέρουν υπηρεσίες σε μη καταγεγραμμένους ε, πρόσφυγες και μετανάστες. Ξεκινώντας από υποψίες, εκφοβισμό, ε, πειθαρχικέ κυρώσεις και καμιά φορά και καθαρή ε, ποινικοποίηση, όπως έχουμε δει και σε περιπτώσεις έρευνας και διάσωσης κατά ορισμένων επιχειρήσεων υπερπροσφύγων. Δεν είναι υποθετική περίπτωση αυτή, είναι προτεραιότητα απέναντι στις προσεγγίσεις ασφάλειας που μπορούν να οδηγήσουν σε καταστάσεις όπου Εδώ λοιπόν βλέπετε αυτούς που λαμβάνουν, χρήσιμα, ε, ε λαμβάνουν χρήματα μάλλον από χρηματοδότηση για θέματα μετανάστευση για την ε, κατασήγηση της κριτικής κατά των ε, κυβερνητικών αρχών. Ορισμένες μάλιστα οργανώσεις αποφεύγουν να παρακολουθούν την πορεία των ανθρώπινων δικαιωμάτων διότι φοβούνται ότι θα χάσουν την η δημόσια χρηματοδότηση χρησιμοποιείται άλλωστε καμιά φορά για να περιορίζονται τομείς δραστηριότητας που δεν είναι δικαιούχοι χρηματοδότηση. Και εκεί υπάρχει η δυνατότητα των χωρών μελών να αποφασίζουν εάν πολίτες, αλλά επίσης και δήμοι, ή βλέπετε ένα γράφημα το οποίο δείχνει πως η χρηματοδότηση είναι και μία από τις ανησυχίες Ιδίω η ανησυχία αυτή είναι υψηλή στην Ιταλία, λιγότερο στην Ουγγαρία. Βέβαια εκεί έχουν άλλε μάλλον είδου ανησυχίες που έχουν άλλη προτεραιότητα και συχνά αμφισβητείται, του έχει ζητηθεί καμιά φορά να, να, δώσουν και τα προσωπικά δεδομένα και να παραδώσουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα των προσώπων στα οποία προσφέρουν υπηρεσίες. Αναγνωρίζουμε ωστόσο του πλαισίου το European Values Instrument είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Πρέπει να τονιστούν εκεί τα ε, σχετικά θέματα και στα πλαίσια της ε, μετανάστευσης και του ασύλου. Το άλλο, Litigation Fund, ταμείο δηλαδή για την επίλυση διαφορών ε, που υποστηρίζει ο δικαίου, μπαίνει ως αιρεσιμότητα στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό το βλέπουμε εμεί θετικά, αλλά δεν θα πρέπει να παραμείνει ε, μόνο θα πρέπει να αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου. Δηλαδή πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιος κάνει τι. Γιατί μπορεί να έχουν διαφορετικές διοντολογίες και διαφορετικούς κανόνες. Ε, υπάρχει και η πολιτική προτεραιότητα για χρηματοδότηση για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και αυτά πρέπει να ε, είναι βέβαια σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα ιδίως για στέγαση, προσφορά ε, τροφίμων κλπ. Είναι σημαντικό επίσης να δημιουργηθεί ένα διαρκές παρατηρητήριο το οποίο θα παρακολουθεί τις, ε, να δοθούν και νέες δυνατότητες στους ε, φορείς κοινωνίας των πολιτών για να υποβάλει καταγγελίες και να κάνει το λεγόμενο shadow reporting. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Uh, Ο τμήματάρχης στην Διεθνή Οργάνωση για Μετανάστευση ε, να πάρει το λόγο για πέντε λεπτά και να μας κάνει μια παρουσίαση. Ή τμήματάρχης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο και συγχαίρω το Κοινοβούλιο που μια εισαγωγή για την επόμενη φάση δηλαδή. Ως ε, οργάνωση για την ε, μετανάστευση θεωρούμε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις για το πουδουπού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά. Πέρασαν τρία χρόνια από τη στιγμή που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση την ατζέντα για τη μετανάστευση μετά την κρίση την ε, μεταναστευτική. Αν δούμε το της μετανάστευσης, αλλά από τους τέσσερις πυλώνες που είχαμε, τώρα έχουμε τρεις μόνο πυλώνες. Γιατί το άσυλο και οι πρόσφυγες έχουν μπει σε ένα πυλώνα της μετανάστευσης, αντί ε, για την τάση για να αξιοποιήσουμε μετανάστευση θα πρέπει να σταματήσει, αν θέλουμε να έχουμε αυτή την πρωτοπόρα θεώρηση για τη μετανάστευση. Ένα από τα πρώτα ε, έγγραφα της Κομισιόν για, την, για το MFF, για το Πουδουπού, λέει ότι θα πρέπει, θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μετανάστευση. Και ο προπολογισμό, επομένω, θα πρέπει να είναι το μέσο για την εφαρμογή αυτού του πράγματο. Επομένω, με τι θα πρέπει να μοιάζει αυτή η στρατηγική. Καταρχάς η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αλλαγή για να αποκτήσουμε νέες φιλοδοξίες για την διαχείριση της μετανάστευσης. Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρχει μια πραγματική συνεργασία και μια πραγματική εταιρική σχέση. Μιλάμε για φτωχέ χώρες με τις οποίες θα πρέπει να συνεργαστεί η Ένωση και θα πρέπει να τι δει κοινά επωφελή ε, διακυβέρνηση της μετανάστευσης. Επίσης θα πρέπει να έχουμε πολιτικές καινοτόμες, ε, συνεκτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να γνωρίσουμε τις τάσεις τις δημογραφικές, της ε, αγοράς εργασίας, δυνατότητες νόμης μετανάστευσης, αλλά και επιστροφής με αξιο άνθρωποι αυτοί που επιστρέφουμε. Και να μην ξεχάσουμε την, ε, τις υποχρεώσεις αλληλεγγύης και διεθνούς προστασίας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάγκη να εξασφαλίσουμε τη συνοχή στο εσωτερικό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά θα πρέπει ούτω ώστε να εφαρμοστεί, να υλοποιηθεί αυτό το όραμα. Το νέο Πουδουπού είναι μια νέα ευκαιρία, ε, γιατί θα γίνουν και παράλληλα συζητήσεις ε, για το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Ε, η χρηματοδότηση της ε, μετανάστευσης θα πρέπει να γίνει με πιο στρατηγικό τρόπο, ούτως ώστε να μεγιστοποιήσουμε, όπως είπαμε και στο παρελθόν, την προστιθέμενη αξιολιστική προσέγγιση, μια ισορροπημένη προσέγγιση και μια απλή προσέγγιση, πραγματικά απλή, ούτως ώστε να μειωθεί και το διοικητικό άχθος για την εφαρμογή της και για να μπορέσουμε να εστιάσουμε εκεί που πρέπει. Περιμένουμε να δούμε τι θα δώσουν οι διαπραγματεύσεις που μόλις ξεκίνησαν με την πρώτη πρόταση που υπέβαλε η Κομισιόν στις 2 Μαΐου. Θα σκεφτούμε λοιπόν και τις συναντήσεις του Συμβουλίου που θα γίνουν στις 28 και 29 Ιουνίου που θα συζητηθούν τα θέματα μετανάστευσης. Ούτως ώστε να γίνει μια υγιή συζήτηση ε, για ένα συνεκτικό όρο από τη μετανάστευση. Because I don't see members of the parliament. την κυρία Γέλα Σέντερ. Έχετε το λόγο. Ήθελα να πω δύο λόγια για αυτό που συνέβη στην παρουσιαφάση. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι η μετανάστευση κατανέμεται και διαιρείται σε διάφορες δραστηριότητες πρόσφυγες και τούντες άσυλο. Να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι μιλάμε για τη μετανάσταση μιλάμε για το θέμα των προσφύγων και μιλάμε και για το θέμα των ε, επιτυχών αιτήσεων για άσυλο. Όλα τα υπόλοιπα δεν περιλαμβάνονται. σε ό,τι αφορά δηλαδή την επιστροφή των ε, προσφ... μεταναστών των άσυλων και των προσφύγων για να μην καταρρεύσει το σύστημα. Να σας ευχαριστήσω γιατί ξέρουμε επακριβώς ε, ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσουν όλα αυτά τα πράγματα επί τόπου χωρίς εσά, γιατί δεν έχει πολύ απλά διαχείριση διαχείρισης Ευρωπαϊκή Ένωση επί τόπου για να επιτελέσει αυτό το έργο της ενσωμάτωσης τη ένταξη Να πω και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξή. Είναι εντελώ απαράδεκτο ότι τρία χρόνια μετά το μεγάλο αυτό κύμα και μετά από τη λειτουργία του ΑΜΕΦ, δεν ξέρουμε ακόμα τι κοστίζει πόσο σε ποιο κράτος μέλος. Έχετε εσείς τέτοια στοιχεία για το τι στοιχίζει η ένταξη, η ενσωμάτωση των προσφύγων στην Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία. Δεν έχουμε αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε πολύ γενικά αριθμητικά στοιχεία και τελικά εξελίξεις τις οποίες δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε. Δεν μπορούμε να κινηθούμε λοιπόν με έναν ε, σωστό συνολικό τρόπο για να ξέρουμε αυτά που κάνουμε αν ε, αρκούν και αν είναι τα σωστά μέτρα. Ήμασταν, μεταβήκαμε στην ε, Ελλάδα, στην Λέσβο, στο Μωρία, στο, Μωρία, στο, προσφυγικό καταβλισμό και για παράδειγμα μας ενημέρωσαν ότι λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τα τρόφιμα. Ρωτήσαμε πόσο κοστίζει λοιπόν ένα γεύμα δεν ξέρω να μας πούν. Δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε λοιπόν τι κάνουμε. Και γι' αυτό λοιπόν, ε, αν θα μπορούσατε να τοποθετηθείτε για όλα αυτά, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την των ε, εμπλεκόμενων φορέων που έγιναν στην ε, μελέτα. Χρειάζεται μια κεντρική αρχή συντονισμού για να συντονισμού και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί με τον τρόπο αυτό η κατάσταση. Δεύτερη ερώτηση. Κάποιοι από τους εμπλεκόμενους φορείς με τους όπους με τις εθνικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη τι θα πρέπει να αλλάξουν για να βελτιώσουν τα εφιστάμενα συστήματα προκειμένου να είναι πιο πέντερ. Σε ευχαριστώ πολύ. Είδα ότι και εσείς είχατε σηκώσει το χέρι και μάλιστα πριν από μένα. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να θέσω κι εγώ ερωτήσεις. Άκουσα με μεγάλη προσοχή αυτό που είπαν οι εκπρόσωποι των διαφόρων πάρα πολύ εμπειρία και που προσπαθούν να μας βοηθήσουν για να επιλύσουμε μία από τις πιο σοβαρές κρίσεις που αντιμετωπίσαμε στην ιστορία μας μαζί με τη δική μας ε, κοινωνικό-οικονομική κρίση, την αμυγός ευρωπαϊκή. Έτσι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι τα πράγματα. Ε, έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ποιες είναι οι βασικές θεμελιώδεις αρχές που κατευθύνουν αυτή την ε, πολιτική. τις οποίες προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Ε, είτε είναι πρόσφυγες ε, λόγω φτώχειας ή κλιματικοί πρόσφυγες ή μετανάστες οι οποίοι απλώς φεύγουν από την πατρίδα τους για να βελτιώσουν την προσωπική τους κατάσταση. Και γι' αυτό έρχονται. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σε επίπεδο πρόληψης και ποσοτικά, δηλαδή να επενδύσουμε τώρα χάρη στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, με ποιο τρόπο Αυτέ οι επενδύσεις. Όταν εγώ πηγαίνω σε διάφορε αποστολέ και έρχομαι σε επαφή με ΜΚΟ, βλέπω ότι παραπονιούνται γιατί ένα τμήμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού επιστρέφει στους εθνικούς προπολογισμού. Παραπονιούνται γι' αυτό. Ορισμένε φορές μας επικρίνουν γιατί ορισμένα προγράμματα Καταρχάς είναι πολύ κατακαιρματισμένα. Α, λεφτά. Δεν φτάνει στα χέρια τους, δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό, δεν τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν αυτά που πρέπει. Δεύτερον, όταν έχουν ξεκινήσει οι μεταναστευτικές ροές, όταν ξεκίνησαν μάλλον οι μεταναστευτικές ροές, ε, εμείς τι κάναμε. Το βασικό είναι να υποδεχτούμε αυτούς τους μετανάστες, αλλά με ασφάλεια. Ε, να μην προωθήσουμε κάποιες μορφές απάνθρωπης μεταχείρισής τους, κλαβιάς και τα λοιπά, να μην συνεχίσουν αυτή η κατάσταση, ας πούμε, στις ακτές της Λιβύης, γιατί μετά δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Πρέπει να διασώσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους ε, επιστρέψουμε πού, σε ποια χώρα ε, τους επιστρέφουμε σε χώρες, ας πούμε αν τους επιστρέφουμε στη Λιβύη, δεν υπάρχει σωστή υποδοχή ούτε καταχώρησή τους. Με ποιον τρόπο λοιπόν θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Μεταναστεύουν. Και για μας φυσικά που τους δεχόμαστε. Και το τελευταίο κομμάτι φυσικά είναι η ένταξη. Είναι το πιο σημαντικό θέμα. Γιατί οι ποσοστώσεις δεν ε, λειτουργήσανε. Ε, Ποια είναι η σημερινή κατάσταση. Ε, κρατάμε. Ε, ενώ έχουμε χώρες όπως η Ουγγαρία, ας πούμε, οι οποίοι λένε όχι στη μετανάστευση και όπου αυξάνεται ο λαϊκισμός. Πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε λοιπόν κάποιους τρόπους, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την ένταξη των ανθρώπων αυτών. Και να δούμε, να μην το κρύψουμε. Υπάρχουν δημοκρατικά προβλήματα στην Ευρώπη. Ε, αυτό συνδέεται και με την οικονομία μας. Αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν εδώ, είναι στη γη μας ε, και όμως δεν τους αξιοποιούμε. Έχουμε λοιπόν αυτά τα βασικά θέματα. Έχουμε το θέμα του προπολογισμού. Ο προπολογισμό. Προωθήσουμε διάφορα προγράμματα με ευρωπαϊκό χρήμα, ευρωπαϊκά κονδύλια, δεν ξέρω πώς. Ε, να αξιοποιήσουμε ήδη αυτά τα προγράμματα που έχουν λειτουργήσει καλά, που είναι επιτυχή. Ε, έχουμε διάφορη εμπειρία από τις χώρες προέλευσης, από τις χώρες διέλευσης και από τις χώρες άφηξης. Πώς μπορούμε κάποιους άξονες ε, συστηματικούς ε, που να είναι υποφελείς για όλα τα κράτη-μέλη. Πριν πω οτιδήποτε, θέλω να σας πω ότι μου φαίνονται εντυπωσιακά αυτός να, προσπά... παρά να προσπάσει πραγματικά ο κ. Λετζέρη να θολώσει τα νερά. Τέλος πάντων, για αυτά που ακούσαμε από τους ομιλητές. Αυτά ήταν πολύ ενδιαφέροντα, πολύ χρήσιμα πιστεύω. Θα ήθελα να ρωτήσω τις οργανώσεις κοινωνία των πολιτών, έτσι με απλά λόγια. Εμείς, μια και έχουμε λόγο στον προϋπολογισμό, ούτως ώστε να μπορέσετε να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας. Μία αλλαγή, πιο σημαντική κάτι γνώμη σας, ποια θα ήταν αυτή. Επίσης, από την ημερήσια διάταξη δεν φαίνεται για το μέλλον τι θα γίνει και ό,τι αφορά την ενσωματώση. Για το μέλλον τι θα γίνει και ό,τι αφορά την ενσωματώση. Παρμογή της ανάθεσης συγκεκριμένων ε, κονδυλίων για συγκεκριμένους ε, σκοπούς. Όλα αυτά είναι υπό εξέλιξη. Δεν μπορώ να απαντήσω.